Bene. Να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα την Επίτροπο Νέλη Κρούς που ήρθε μαζί μας εδώ. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αρμοδιότητα τους τομείς ε, και τον διελθωμένο διάλογο, τους τομείς του, των αρμοδιοτήτων της και τον διελθωμένο διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο. Να ξεκινήσουμε αμέσως, για να γίνει συζήτηση μετά, θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην Επίτροπο για την εισηγησή της. Thank you. Uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει η Επίτροπος. Είναι μεγάλη μου χαρά. Εδώ να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Μια που έχουμε καλύψει σχεδόν τη μισή περίοδο για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι όσον αφορά την περίοδο αυτή, αυτή μες στη θητεία. Μας μείνει ακόμα ένας χρόνος και κάτι μήνε, ακόμα έχουμε πολλή δουλειά και εγώ είμαι αποφασισμένη να συνεχίσουμε την ίδια όρμη και ενέργεια, οπότε επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να σα μιλήσω, να σα πω τι γίνεται όσον αφορά το διαδίκτυο, όσον αφορά το ανοιχτό πνεύμα, ανοιχτή φιλοσοφία και κάποιε ευκαιρίε και την καινοτομία. Αυτά, αυτά είναι τα θέματα για τα οποία πρόκειται να σα μιλήσω. Επίση να σα πω και άλλα δύο λόγια για την ενιαία αγορά για την επικοινωνία, ας πούμε. Και να πούμε και δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο της περασμένης εβδομάδας. Πρώτα από αυτό το ανοιχτό πνεύμα, ανοιχτή φιλοσοφία, το διαδίκτυο. Έτσι είναι, μια ανοιχτή πόρτα. Είναι μια πλατφόρμα παραγωγική, ε, ισχυρή και αυτό διότι είναι ανοιχτό, οπότε θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτή την ισχύ του Ιντερνετ με το ανοιχτό πνεύμα και Επομένω θα πρέπει και οι κανόνε του οποίου έχουμε θέσει να ανταποκρίνονται, να αντιστοιχούν σε αυτό το ανοιχτό πνεύμα και επομένω να καταργούν φραγμού, εμπόδια και θα πρέπει να δημιουργούμε οικονομίε κλίμακα. Να σα πω πώ τα κάνουμε όλα αυτά. Πρώτα-πρώτα το, το, το σύννεφο. Οι επιχειρήσει, οι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτε, θα πρέπει να προσφέρουν ε, τεχνολογία, πιο φθηνή και για τους ε, πολίτες και για τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να, ε, το για τον πολίτη να είναι τελικά κάτι σαν ένα, ένα ντουλεπάκι ερμάριο το οποίο να είναι επιγραμμικό να, ε, για την αγαπημένη μουσική, βιβλία κάποιου και θα πρέπει βέβαια να μην υπάρχει κατάτμιση της αγοράς από τους κανόνες. Και αφού μιλάμε για κοινή αγορά θα πρέπει να μιλάμε και για κοινά στάνταρ, κοινά πρότυπα, αλλιώς δεν είναι εκείνη αυτή η αγορά. Και περιμένω πώς και πώς να λάβω γνώση της έκθεσης της Πιλάρ del για τη στρατηγική που αφορά το σύννεφο του, αυτό το cloud. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το copyright, για δημοτικά δικαιώματα, γιατί πρόκειται για ε, έναν τομέα που επιδέχεται αλλαγές. Εδώ και πάρα πολύ καιρό απαιτούνται και αλλαγές και η ε, εξής τεχνολογίας μας έχει οδηγήσει και σε αυτόν τον τομέα στην ανάγκη για αλλαγές. Οπότε τώρα θα σας πω ότι κάποιοι ονομάζουν ότι δεν μπορούμε με νόμιμο τρόπο να έχουμε πρόσβαση σε ταινίες, σε μουσική, και ε, οι τέλτες λένε δεν μπορούμε να, να, να τον κόσμο που θα θέλαμε, ε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι τεχνικέ λένε οι επιστήμονες, όμως υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει αναλεκτική εναλλακτική ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το κόπηρα το σχετικό δίκαιο και οπότε τότε θα ικανοποιήσουμε περισσότερου ε, και τον κόσμο και του καλλιτέχνε και του επιστήμονε. Και κυρία Πρόεδρε, γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή την υπόθεση που λέγεται Licenses for Europe, ε, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις για την Ευρώπη και ε, δεν, δεν, δεν είμαι τόσο θαυμαστής της νομοθεσίας, αλλά πρέπει να, είμαστε ρεαλιστές και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες λύσεις οι οποίες να είναι ευκολότερες και λιγότερο γραφειοκρατικές. Ε, Επομένω θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε εξυγχρονισμό με την νομοθεσία. θα πρέπει να γίνει αυτό αφού δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας αλλιώς. Και Επίσης, θα τον ανοιχτό πνεύμα να πρετανεύει και αλλού. Ε, ας πούμε στην ενημέρωση του κόσμου θα πρέπει επομένω οι δημόσίε υπηρεσίε, η διοίκηση να διακρίνεται περισσότερη διαφάνεια να υπάρχουν προϊόντα και υπηρεσίες που να σχετίζονται με την, την αξιοποίηση των δεδομένων και επίση θα πρέπει έτσι να βοηθάμε να δίνουμε όθηση στην αγορά. Γιατί μιλάμε εδώ πέρα για δεκάδες δι ευρώ και πάρα πολύ σωστό ε, ότι τελικά νομίζω ότι ο κ. Κάλφεν και οι άλλοι θα κάνουν καλή δουλειά του. Ευχαριστώ. Ελπίζω τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία φιλόδοξη πριν κλείσει η Ιρλανδική Προεδρία. Οπότε όλοι να μπορούν να έχουν ε, να χρησιμοποιούν και να επαναχρησιμοποιούν παρακάτω αυτού του είδους τα δημόσια δεδομένα και επομένως να υπάρχει αξία, προστιθέμενη αξία η οποία να παράγεται και να αναπαράγεται σε όλη την αγορά και οπότε δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει, να παραλείψει αυτό το πνεύμα ελευθερίας, το την ανοιχτή φιλοσοφία που εξαρτάται και από την ασφάλεια. Αλλιώς κανένας ε, κινδυνεύει να, να υποστεί υπεξαίρεση ταυτότητας, ε, να τον κατασκοπεύσουν, ε, να τον μολύνουμε Ιού πλήρω και οπότε γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι να έχουν ανοιχτό πνεύμα ε, και να ανοίξει ο τομέας αυτό για τις υπηρεσίες όλη είναι η αγορά, γι' αυτό χρειάζεται κυβερνοασφάλεια, έχουμε τη σχετική οδηγία και θα πρέπει να είναι και ανθεκτικά τα δίκτυα, γιατί οι απειλέ που προανέφερα δεν γνωρίζουν σύνορα για να τι αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Και γι' αυτό και σα λέω, κυρία Πρόεδρε, ότι με μεγάλη μου χαρά παρουσιάζω τη σχετική στρατηγική το Φεβρουάριο. Political priority Μιλάμε για κάποια υψίστη προτεραιότητα. Για όλους πολιτική προτεραιότητα και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να κάνει γοργά βήματα προόδου και έτσι η οδηγία για τη δίκτυα και για την ασφάλεια της πληροφορίας θα εγκριθεί κατά αυτή τη θητεία. Και αυτού του είδους η ελευθερία, ε, αυτού του είδους το ανοιχτό πνεύμα αφορά την ίδια αγορά, ε, όλα γίνονται ψηφιακά, έχουμε επιλογή. Θα συνεχίσουμε μέσα να έχουμε όμως φραγμούς όσον αφορά το, το, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την καινοτομία. Ε, επί δεκαετίες καταρρίξαμε τους φραγμούς σε άλλους τομείς, οπότε και τώρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε την νέα αγορά, η οποία να είναι ζωντανή, να έχει ενέργεια, να είναι ενωμένη, να είναι ανοιχτή και αυτό έχει σημασία και εκτός της ενιαία αγοράς, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις, τις αρετές, τα πλεονεκτήματα, την αξία αυτή ε, αυτής της και αναγνωρίζουμε επομένω το ότι τα ωφέλη δεν είναι μόνο οικονομικά, αφορούν και την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατία. Οπότε, ε, βέβαια, δεν ισχύουν αυτές οι αξίες παντού. Σε όλες τις χώρες και έχουμε διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε διεθνείς συναντήσεις παντού. Από το IGF του Μπακού μέχρι το WCIT στο Ντουμπάι. Ας προσπαθήσουμε αυτό το χάσμα να το γεφυρώσουμε όταν, όπου είναι δυνατόν, ας προσπαθήσουμε να μην περιθωριοποιούμε κανένα και να βοηθούμε στη δημιουργία δυνατοτήτων. Όμως τελικά μερικοί θέλουν περισσότερο κυβερνητικό έλεγχο. Εάν αυτοί κερδίσουν το παιχνίδι, τότε ποιο είναι ο κίνδυνος ότι θα έχουμε κατάτμιση του διαδικτύου. Οπότε θα χαθούν τα πλεονεκτήματα του ενιαίου παγκόσμιου ανοιχτού ε, δικτύου. Και γι' αυτό και συνεχίζουμε και προωθούμε τις αξίες Ευρωπαϊκής συνεχίζουμε να θέλουμε ε, ένα ανοιχτό μοντέλο που να έχουν πολλούς εμπλεκόμενους και αυτό να είναι το πρότυπο για τη ε, διαδικτυακή διακυβέρνηση οπότε ας ακουστεί ενιαία φωνή από την Ευρωπαϊκή Ένωση σωστή εκπροσώπηση προς τα έξω, κοινή γραμμή και υπέρ του να έχουμε ένα ελεύθερο και εύρο στο Ιντερνετ. Τώρα, το δεύτερο που θέλω να σα πω είναι το εξή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό ο ψηφιακό μετασχηματισμό προσφέρει μια ευκαιρία για όλου του συμπολίτε μα. Διότι χρειάζεται εδώ πέρα κάποιο είδου αυτοπεποίθηση ψηφιακή, κάποιου δεξιότητε. Πολύ σημαντικά. Ε, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο που θα θέλαμε, γιατί σύντομα ίσω θα έχουμε ε, έλλειψη ε, σχεδόν ενός εκατομμυρίου εξειδικευμένων ε, τεχνικών, επιστημών, τεχνοκρατών ε, στην ε, τεχνολογία των υπολογιστών και οπότε αυτό είναι τρελό, είναι παράλογο μια που υπάρχει τόση ανεργία γύρω γύρω άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ευρυσκοτά μας είναι τρομερό αυτό και τα κρατημέλη νομίζω ότι πασχίζουν να δουν τι θα γίνει έχουμε αυτό το 60-50% που έχουμε φτάσει σε ε, νέων, Απαράδειγη κατάσταση. Επομένω αν θα μπορούσαμε να συγκεράσουμε αυτού του δύο στόχου λίγο περισσότερο, σε αυτή την περίπτωση θα βοηθούσαμε, θα βοηθούσαμε την νεολαία. Αλλά θα κάνουμε και βήματα προόδου στην ανταγωνιστικότητα. Πάντω μπορούμε κάτι να κάνουμε για να άρουμε αυτό το κενό που υπάρχει την έλλειψη από πλευρά τη βιομηχανία, από πλευρά τη εκπαίδευση, γιατί ε, όλοι μα έχουμε δεσμευτεί να προσπαθήσουμε αυτή την και έχουμε κάνει deal με, με τους ε, συνεταίρους μας και έχουμε αυτή τη, μεγάλη συμμαχία για ψηφιακές θέσεις Χρειάζεται επομένω μια καινούργια συνεργασία ώστε να, μπορέσουμε να θεραπεύσουμε ε, ε, τα, τα προβλήματα της οικονομίας και δεν χρειάζονται λόγια, αλλά χρειάζεται δράση, χρειάζονται δεσμεύσεις, όχι μόνο την Κομισιόν, αλλά από όλους. Ε, όλοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και θα πρέπει να βρεθεί μια νέα εταιρική σχέση. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν περιθωριοποιούμε το μισό κόσμο. Ε, η σταδιοδρομία στην τομέα της πληροφορικής δεν ελκύει αρκετά τις γυναίκες ή αρκετές γυναίκες, διότι οι γυναίκε, οι νέε γυναίκε τέλο πάντων, θεωρούν ότι δεν είναι για εκείνε η τεχνολογία των υπολογιστών. Ε, κάνουν λάθο. Όλοι μπορούν να έχουν προσβασιμότητα εκεί και είναι μια ευκαιρία για όλου. Και θεωρώ ότι είναι υπέροχο το ότι συνεργαζόμαστε όσον αφορά την ημερίδα εκείνη που ονομάζεται νέε κορίτσια, νέε γυναίκε και τεχνολογία υπολογιστών. We also need to focus on innovation. Um, so much of επομένω να έχουμε καινοτομία και η καινοτομία αυτή φυσικά και μπορεί να προέλθει από του επιχειρηματίε, οπότε ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε οι περισσότερε εταιρείε τη απασχόληση έρχονται από εταιρείε που μόλι ανοίγουν και πολλέ φορέ πρόκειται για διαδικτυακέ επιχειρήσει. Όμω αυτό θα πρέπει να το μεταλαμπαδεύσουμε και εδώ και θέλουμε να υπάρχει τέτοιου κουλτούρα που αμείβει τον επιχειρηματία. Αλλιώ ρισκάρουμε την αποτυχία και εν πάση περιπτώσει θέλουμε να υπάρξει σωστή υποστήριξη, ή πόροι για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία για καινούργιε εταιρείε, για καινοτόμου, για ερευνητέ και έτσι να ωφεληθούν οι νέοι. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά που γίνεται. Ξεκίνησε αυτό στην Ισπανία με την τηλεφώνικα και στο Βερολίνο 10.000 Ναι, το καλοκαίρι. Εκεί είναι πλάκισμα και το καλοκαίρι αυτό το κάμπους αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο Λονδίνο. Να, πώ δημιουργούνται τα πράγματα, και Επίσης, με θεωρώ ότι είναι υπέροχο ότι ο κοινωνικός προπολογισμός θα συνεχίσει να στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία. Το Δεορίζον 2020 είναι μια όθεση πιο μεγάλη από ποτέ για την οικονομία. Και επομένω, η πληροφορική μπορεί εδώ πέρα να βοηθήσει πάρα πολύ με κάποιους απλούς κανόνες, έτσι μπορούμε να ε, το κάνουμε ευκολότερο για τις περισσότερες ε, καινοτόμε εταιρείε, να καλυφθούν ε, με, χρηματοδότηση, να δώσουν περισσότερο προϊόντα στην αγορά, να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα από το ορίζον 2020. Νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσει να την προσοχή μας σε τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρονικά, η ηλεκτρονική τελος πάντων και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά συστατικά αυτού του οικοσυστήματος και να δούμε πως δεν θα έχουμε κατάτμιση, δηλαδή να έχουμε ένα έρμπας από κάποια μικροκυκλώματα τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αρένα. Ε, τέτοιου είδου καινοτομία επομένω μπορεί να δώσει όθηση και να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις αύριο. Αυτό, αυτό είναι το όνειρό μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα υπερταχαία δίκτυα, γιατί εδώ για 10 χρόνια έχουμε ε, τις ε, που θα αυξηθούν 33 ε, φορές. Οπότε πάμε τώρα για τεχνολογία πέμπτης γενιάς. Όμως ε, αυτή η τεχνολογία πρόκειται να φτάσει στο να φτάσει και να ξεκινήσει από την βιομηχανία της Ευρώπης με ευρωπαϊκή έρευνα κλπ. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να έχουμε συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Να μπορέσουμε να γίνουμε ξανά πρωτοπόροι όσον αφορά τεχνολογία. Αυτό θα τονωθεί με επενδύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίω όλα αυτά, η ελευθερία, οι ευκαιρίε, η κοινοτομία, όλα αυτά εξαρτώνται από τι, από την ευρυζωνικότητα, διότι οι Ευρωπαίοι νοιάζονται για το ίντερνετ. Κάνουν ουρέ έξω από τα καταστήματα για να αγοράσουν την τελευταία συσκευή, τελευταίο gadget και διαμαρτύρονται για τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται στο διαδικτυακό περιεχόμενο όμως ε, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία χωρίς την ευρυζωνικότητα, τα ευρυζωνικά δίκτυα. Οπότε θέλουμε να υπάρχει, να ισχύσει τέλο πάντων αυτό μας το πρόγραμμα, το σχέδιο, το πρόγραμμα των 10 σημείων για την ευζωνικότητα. Και έτσι να φτάσει όλη η ευζωνικότητα. Όμω, το Συμβούλιο το κολόβωσε αυτό το πρόγραμμα, το περιέκοψε όσον αφορά αυτού του είδου την ε, Connecting Europe Facility όπω ονομάζεται και εγώ είμαι όμω αποφασισμένη, θα χρησιμοποιήσω κάθε κονδύλιο στο οποίο έχω πρόσβαση. Από την ΕΤΕ, από το, το Ταμείο Επενδύσεων, το Διαρθωτικά Ταμεία, από παντού. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σα, ώστε αυτό το μήνυμα να φτάσει στου συναδέλφου σα στην Περιφερειακή Επιτροπή και Επιτροπή των Προπολογισμών. Γιατί είδαμε τι έγινε στο Συμβούλιο, τι έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτε. Δεν άδρεξαν την ευκαιρία, τη χάσανε. Πάντω, ειλικρινά, ελπίζω ότι εσεί, το Κοινοβούλιο, Κάνετε διόρθωση πορείας. Βεβαίω. εγκρίνουμε και άλλα μέτρα για τις ε, γενικές υπηρεσίες και για την ε, καθολικές υπηρεσίε και για την ουδετερότητα του δικτύου. Την επόμενη εβδομάδα δε πρόκειται να δημοσιεύσουμε την πρότασή μα όσον αφορά την περικοπή των δαπανών για την ανάπτυξη τη ευρυζωνικότητα. Και έτσι, με την χρήση τη ενιαία ε, αγορά, μπορούμε να πετύχουμε για πάρα πολλού κλάδου οικονομίε κλίμακα. Ανά ομάδα συμφερόντων, ανά χώρα να κάνουμε βήματα πρόοδο και δεν είναι δυνατόν να προσκολόμεθα σε κάποιου είδου ε, νομοθετικέ ρυθμίσει και κάποιου είδου ιστορικά δικαιώματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται και επιγόντω είναι μια προσέγγιση η οποία να είναι φιλόδοξη, πραγματικά ευρωπαϊκή. Και αυτή τη φιλοσοφία θα διέπει το, το ε, πρόγραμμα δράσεις το οποίο έχουμε εκπονήσει. Αυτά είναι απλώ η αρχή. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει την ε, αγορά των τηλεπικοινωνιών. Την περσμένη εβδομάδα ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ε, συνάντηση του Οκτωβρίου όσον αφορά την, τους, τους ε, την πληροφορική. Μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, καταλαβαίνετε σήμερα. Θα θέλουμε να μπορέσουμε στις τηλεπικοινωνίες, στα ψηφιακά, να γκρεμίσουν τα σύνορα, και έτσι να μπορέσει η Ευρώπη να είναι ε, ανταγωνιστική παγκόσμια. Θέλουμε επομένως καλύτερες συμφωνίες για τους ανταγωνιστές, περισσότερη ολοκλήρωση, καινοτομία, συνδέσεις, ανταγωνισμό, περισσότερη επιλογή και όλα αυτά επιτέλους ε, ελπίζω να υλοποιηθούν και όσον αφορά τη, την περιαγωγή για όλη την Ευρώπη, οπότε νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να τονώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία κατά 110 ευρώ ετησίως. Ετησίω. Αυτό τι είναι, το 0,8% του ΑΕΠ. Αυτό θα μας απασχολήσει σαν προτεραιότητα τους ε, μέσω επόμενους μήνες. Σε αυτή την καυτή επικαιρότητα που αφορά την απασχόληση. Ελπίζω ότι και εσείς θα παίξετε κομβικό ρόλο σε αυτή την προβληματική. Και περιμένω πώ και πώ τη δική σα ενεργή συμμετοχή. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία του, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια βιζονικότητα για όλου. Και έτσι να εξασφαλίσουμε μια, μια Ευρώπη που είναι ανταγωνιστική, που να είναι συνδεδεμένη. Αυτά θα να σα πω. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε όχι μόνο πλέον για την παρουσία σας, αλλά και για την εισήγησή σας, που από ό,τι βλέπω έχει πυροδοτήσει αλλεπάλληλες, αιτήματα για να λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι. Θέλω να σας ζητήσω όμως μια χάρη, συνάδελφοι. Ο κύριος Φανίστερ Ρόι πρέπει οπωσδήποτε να φύγει στις 4 και θα κάνουμε μια εξαίρεση, θα του δώσουμε πρώτα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να δράξω το, το πλωμένο χέρι της κυρίας Επιτρόπου που ζήτησε να σκεφτούμε δημιουργικά και βεβαίως έχει δώσει το καλό παράδειγμα σε πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες ε, για την εκμετάλλευση των διαφόρων ευκαιριών που υπάρχουν σε καιρούς ε, κρίσης. Κοιτάξτε, εγώ είμαι και εισηγητής για το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εκεί πέρα ρωτάμε το πώς ε, θα μπορέσει ο τομέας της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών να αποτελέσει ένα τομέα προτεραιότητας, ε, έναν τέταρτο τομέα προτεραιότητα, δηλαδή με γύρω στα 80 εκατομμύρια. Και βεβαίω γιατί αισθανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για το μέλλον και για τις δουλειές των νέων ανθρώπων. Δεύτερη παρατήρηση Έχουμε την εντολή ε, διαπραγμάτευσης ε, για ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Εκεί πέρα υπάρχει ένας τομέας ε, τομέας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και το θέμα είναι ακριβώς πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτό με τις πρωτοβουλίες που αναφέρατε. Και με αυτή την οπτική ε, και εγώ μαζί σας εκφράζω τη λύπη μου για το ότι το Συμβούλιο δεν έθεσε ανάλογες προτεραιότητες και εμείς ως Κοινοβούλιο λέμε πως θα πρέπει να έχουμε μια κοινή τέτοια ατζέντα, ένα κοινό τέτοιο πρόγραμμα. Να μας είχατε δώσει τότε, θυμάμαι, ε, μια πλαστικοποιημένη κάρτα που... Τι την έχω ακόμα και λέγατε πως η ευρυζωνικότητα είναι κάτι το απαραίτητο για την νέα περίοδο. Και πως στην Ήπεθρο υπάρχει ακριβώς ένα μεγάλο κενό ευρυζωνικότητας και είναι μια κοινή μας ευθύνη. Λοιπόν, εγώ σας στηρίζω πλήρως. Ευχαριστούμε κύριε Φανίστεροι και για αυτήν την πολύ σημαντική διευκρίνηση και τώρα η κυρία Ντελκαστήγιο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε. Στην αρχή είπατε ότι έχουμε ακόμα χρόνο για αυτή τη θητεία. Ε, όχι, δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι, ότι, ότι τελειώνει η θητεία. νομοθετικά και νομοπαρασκευαστικά μετά το καλοκαίρι στην πράξη λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πάντως σίγουρα μπορούμε να έχουμε όραμα για το τι θα γίνει. Και ο απολογισμό τη θητεία για το δικό σας χαρτοφυλάκιο είναι πάρα πολύ θετικό. Νομίζω ότι πάρα πολύ καλά δείξε το δρόμο για το πού μπορούμε να πάμε, τι θα γίνει με τους διάφορους κλάδους, πώς μπορούμε να δώσουμε δυναμισμό στις οικονομίες, τι να κάνουμε την ανταγωνιστικότητα. Να, επομένως, αυτή σας η μεγάλη συμβολή όσον αφορά το προσανατολισμό, τη διαχείριση που γίνεται για κάθε ένα από αυτά τα μέτωπα. Θέλω να θίξω τρία διαφορετικά ζητήματα. Πρώτα-πρώτα. Τι είπε το Συμβούλιο. Ότι θα πρέπει να προτείνει η Κομισιόν μέτρα κλπ. Για τις επικοινωνίες, για την ενιαία αγορά. Για πέστε μας. Τι είδους μέτρα, προτάσεις, δράσεις θα προτείνετε για να ανταποκριθείτε σε αυτό το οποίο σας ζήτησε το Συμβούλιο. Δεύτερον, σε σχέση με αυτά που είπατε για το ευζωνικό φάσμα, με τη διαχείρισή του, τους διαγωνισμούς, τις προμήθειες, πέρα από την εθνική νομοθεσία. Τι άλλο μπορεί να γίνει σε αυτή μου τρίτον. Γι' αυτό το, το περίφημο, την περίφημη ευρωπαϊκή διευκόλυνση του κύριου Φασίλητη από πλευρά δημοσιονομική, μάλλον δεν προσεχθήκε το θέμα. Τι λέτε να κάνετε. Τελευταίο δε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό για την Ευρώπη. Να δούμε. Τι θα γίνει με τη μετάβαση από την αναλογική τεχνολογία στην ε, ψηφιακή απλευράση κράτους δημοσίων υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ ε, κρίσιμο αυτό. Πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση. Και επομένω θα πρέπει με αποφασιστικότητα να πιάσουν τα πρωταγιάρδα, ώστε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η πορεία αυτή την επομένη θητεία. Ευχαριστούμε, Πιλάρ. Και τώρα, κυρία Σικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο που ήρθε σήμερα εδώ και να την συγχαρώ ξανά επειδή προώθησε αυτή την πρωτοβουλία για τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να προωθηθεί. Μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που ω τώρα δεν έχει γίνει επαρκώ. Ειδικώ σε ό,τι αφορά τι νεαρέ κοπέλε, Ο τομέας τεχνολογίας, των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορικής είναι ένας τομέας που μπορεί να δημιουργήσει πολλέ θέσει εργασία. Θέλω λοιπόν εδώ να σας ενημερώσω και να σας βεβαιώσω ότι σας στηρίζει και το Κοινοβούλιο εδώ. Θα θέλαμε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουμε τις περικοπές ε, στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε αυτό το τομέα για την ερχόμενη επταετία. Ιδίω για το Connecting Europe Facility, για την διευκόλυνση διασύνδεση τη Ευρώπη. Εδώ πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυγχρονίσουμε τις απόψεις της κοινωνίας σχετικά και γιατί πολλά εξαρτώνται από την πληροφορική, τις επικοινωνίες και την τεχνολογία. Ήθελα λοιπόν να γνωρίζετε ότι σας στηρίζει το Κοινοβούλιο στην ε, απόρριψη των προτινόμενων περικοπών σε τομεί που μπορεί να μα δώσουν θέσει εργασία. Επίση, θέλω να κάνω κάποιε ερωτήσει για αρκετέ πρωτοβουλίε που εμφανίζονται στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ αναφέρομαι στην ε, διευκόλυνση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το invoicing. Αυτό θα το δούμε το δεύτερο εξάμεινο της φετινής χρονιάς και πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τον τομέα των δημόσιων διαγωνισμών, των προμηθειών. Μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη τον ε, τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό νέφος και τη σχετική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήθελα να ξέρω πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας υποβάλει κάποια πρόταση σε σχέση με αυτή τη στρατηγική. Βλέπω ότι το περιμένει ο κλάδος αυτό, το ίδιο και εμείς. Οπότε μας ενδιαφέρει το πότε η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να προχωρήσει. Το κατά πόσο θα υπάρχει επίσης μια γενική συμφωνία. Σημειώνω ότι θέλετε να μειωθεί το κόστος της ευρυζωνικότητας και ως προς τις ε, υποδομές και ως προς την διάδοση και το τι θα γίνει με την ηλεκτρονική αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Νομίζω είναι σημαντικές οι πρωτοβουλίες αυτές και τις ε, αναμένουμε διακάως. Πότε θα μας τις υποβάλει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν έχουμε πλέον πολύ χρόνο. Προκειμένου όλα αυτά να ολοκληρωθούν εντό τη θητεία μα, θα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα σχετικέ κινήσει. Έπειτα, τι μέτρα θα προτείνετε να λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο, διότι το Κοινοβούλιο θέλει να σας στηρίξει και νομίζω ότι μπορούμε μαζί να προτείνουμε μέτρα τα οποία να οδηγήσουν στην ανάπτυξη του σχετικού κλάδου στην Ευρώπη και τη ίδια τη κοινωνία τη Ευρώπη. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συμφωνώ πρώτα-πρώτα για τις ανησυχίες των συναδέλφων για αυτές τις περικοπές που θέλει το Συμβούλιο. Εάν περάσει αυτή η πρόταση θα τεθεί εν κινδύνο η ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό όραμα, όπως επίσης και το, το, το, το πρόγραμμα αυτό για το νέφος, το cloud κλπ. Βεβαίω και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον τον ορίζοντα 2020 σε σχέση με το ετεροζωνικό φάσμα. Να δούμε πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα το ψηφιακό σε σχέση με τις τριπικοινωνίες. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε τον κόσμο, τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση με την ψηφιακή τεχνολογία, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πια για τον εξυγχρονισμό της οικονομίας στην Ευρώπη. Να δούμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε επομένω το πλονέκτημα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό με τέτοιες περικοπές του προπολογισμού. Βεβαίω, υπάρχουν κάποια ζητήματα όπως είπατε και εσείς στη συνέργεια των διορθωτικών ταμείων αλλά όλα θα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της συνοχής και συμφωνούμε ότι ο ιδιωτικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις ε, υποδομές που θέλουμε να φτιάξουμε. Και έτσι με κάποιο τρόπο να ελκύσουμε και τις επενδύσεις των ιδιωτών. Όμως με αυτά που είπε το Συμβούλιο, πού να ελκύσουμε κανέναν με τέτοιες περικοπές. Ε, τέλος πάντων, όπως είπαμε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η ευρυζωνικότητα. Χρειάζεται επομένως και απαιτείται ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο να ορίζονται εκεί υποχρεώσεις και δικαιώματα όλων. Για πέστε μας. Πότε θα έχουμε την οριστική πρόταση κανονισμού για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τους σχετικούς διαγωνισμούς. Τη σήμερα ημέρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πάντως να είμαστε ενωμένοι για να πετύχουμε τη σωστή, την κατάλληλη χρηματοδότηση. Εστέ σίγουροι μπορείτε να υπολογίζετε στην Επιτροπή μας, στη βοήθειά της και στη δική μας πολιτική ομάδα, γιατί ακριβώς νομίζουμε πάρα πολύ ότι ό,τι κάνουμε σήμερα και ότι ε, λήψεις πάνω στις επενδύσεις χρηματοδότης θα έχει σοβαρές εμπειρία αύριο. Ευχαριστούμε κυρία Τόμψεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι ήρθατε εδώ πέρα σήμερα γιατί πολλοί από εμά ε, σοκαριστήκαμε όταν είδαμε τον προπολογισμό που πρότεινε το Συμβούλιο. Ήταν απίστευτο ότι περιεκόπη η ευρυζωνικότητα κατά 90% και ειδικά μάλιστα λεφτά που είχαν αφιερωθεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Ξέρω πως λέγατε πως η ευρυζωνικότητα ήταν ψηφιακό οξυγόνο για την Ευρώπη γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πού θα βρούμε τα λεφτά. Είπατε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά δεν υπάρχουν παντού διαρθρωτικά ταμεία και κάνατε και κάποιες άλλες προτάσεις. Πότε θα ξέρουμε όμως τι θα υποκαταστήσει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν ελάβαμε. Γιατί πρόκειται για προϋπόθεση για την ψηφιακή Ευρώπη και για τις ε, θέσεις εργασίας που αναφέρατε. Τούτου λεχθέντος για την ευρυζωνικότητα είμαι πεπισμένη πως το Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει και θα το παρακολουθούμε γιατί και οι ψηφοφόροι μας θα τα παρακολουθούν. Επίσης, απομακρυσμένες περιοχές δεν μπορούν να κατοικηθούν γιατί ο κόσμος δεν θέλει να πάει να ζήσει όσο δεν υπάρχει ευρυζωνικότητα. Οπότε είναι ε, σημαντική αυτή η στρατηγική. Δεύτερον, καλά είναι να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, αλλά εκτιμώ πως ε, ο μισός ευρωπαϊκός πληθυσμός ε, δεν ξέρει πώς να ανοίξει έναν υπολογιστή και πώς μπορούμε να διδάξουμε τον κόσμο που φοβάται τους υπολογιστές ε, δεν έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Νομίζω πως θα πρέπει στο κοινωνικό ταμείο κάπου για να υπάρξει μια τέτοια εκπαίδευση. Κοιτάξτε, στη χώρα μου το 2015 θα ψηφιοποιηθεί τελείως το δημόσιο. Και δεν, ε, ο μισός πληθυσμός δεν έχει ιδέα ε, για την πληροφορική. Πρέπει λοιπόν να το πάρουμε σοβαρά αυτό το θέμα. Αλλιώς ε, ο κόσμος θα είναι θυμωμένος. Τέλος θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο είπατε για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Η πιο διαχωρισμένη με βάση το φύλλο αγορά εργασίας είναι αυτή της πληροφορικής και στα πανεπιστήμια δεν, ε, στο δυτικό κόσμο δεν ε, υπάρχουν σχεδόν καθόλου γυναίκες ε, στα τμήματα πληροφορικής πλην Ρουμανίας, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να προσελκύσουμε λοιπόν τους πιο ταλαντούχους και οι επιχειρήσεις. Γιατί είναι ικανοποιημένες με το να επιλέγουν από το 48% του πληθυσμού. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια, ειδικά όταν λέτε πως ε, υπάρχουν ένα εκατομμύριο τέτοιες εργασίες κενές, πρέπει να προσελκύσουμε κορίτσια σε αυτό το κλάδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Μαρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κυρία Επίτροπε, στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε. Θα ήθελα να σχολιάσω την πληροφορική και τον ορίζοντα 2020 και τα σχετικά αιτήματα. Όπως ξέρετε, πληροφορική και τηλεπικοινωνία είναι στον πυλώνα 2, κάτι το οποίο δηλαδή είναι εγκάρσιο σε όλους τους ε, πυλώνες ε, βιομηχανία, ανταγωνιστικότητα, κοινωνικές αλλαγές και τα λοιπά. Όμως, υπάρχει το σχετικό ε, έργο για το, το ΦΑΤ, το λεγόμενο, το οποίο θέλουμε να το προωθήσουμε και στην τεχνολογία και τις ε, θετικές επιστήμες. Οπότε θα θέλαμε την στήριξή σας για την διεύρυνση και την εμπάθυνση αυτού του έργου. Κατόπιν ε, ανοιχτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, κατά το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα. Αλλά ε, ζητάμε από την Κομισιόν με ποιον τρόπο θα υπάρξει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο εντό του ορίζοντα 2020, τη στρατηγική δηλαδή για τι δημοσιεύσει, για να διασφαλίσουμε πώ θα έχουμε πρόσβαση, όπω είπα, αλλά να βελτιωθεί και το επίπεδο πρόσβαση και να προσελκύσουμε και του καλύτερου τους να θέλουν δηλαδή να δημοσιεύουν στα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά και να μην ε, αποθούνται από το ότι δεν έχουμε ε, μια ανοιχτή πολιτική δημοσίευση. Γι' αυτό χρειάζεται ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για να υπάρχει αυτή η πρόσβαση. για να προωθήσουμε τη στρατηγική 2020. thank you, Commissioner, for being here. I... Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Έλερ. Κυρία Επίτροπε, θέλω να τονίσω πως δεν πρέπει ε, μόνο να αναφέρουμε τα αρνητικά της απόφασης του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο έχει οριστεί είναι το πλαφόν. Τι κάνει το Κοινοβούλιο. Ε, δεχόμαστε το πλαφόν. Πέρα από αυτό δεν έχει κρυφθεί τίποτα άλλο. Ειδικά αν δείτε το πώ έχει οικοδομηθεί το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη, το έχουν σπάσει στα δύο και μετά βάζουν μέσα τα διαρθρωτικά ταμείο, ταμεία. Αλλά μετά μειώνουν την ευρυζωνικότητα στο ελάχιστο, το στο ένα δισεκατομμύριο, αλλά δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά αλλού. Οπότε στο πλαίσιο της εντολής ε, του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο μπορεί να το αλλάξει αυτό. Οπότε δεν είναι μόνο ζήτημα του πώς μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο το Συμβούλιο. Πρακτικά νομίζω πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις, γιατί αυτό το οποίο μας προσέφερε το Συμβούλιο ήταν μια κάποια ευελιξία. Και βεβαίως το ζήτημα ήταν το ότι με την ε, διαφορετική αυτή θα δημιουργηθεί κάποιο είδους ε, ταμείο και θα έχουμε κάπου μεταξύ 35, 30 και 45 δισεκατομμυρίων. Οπότε δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το ποσό, ε, γιατί αυτό θα ήταν ε, κάποια εικασία, αλλά με την δέσμευση των χρημάτων. Οπότε το ζήτημα είναι πως θα υπήρχε μια διαφορετική ισορροπία στο πλαίσιο του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, γιατί θα χρησιμοποιούσαμε κάτι από τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεύτερον, μπορούσαμε στο πλαίσιο ποσοστών να κατανείμουμε τα λεφτά εντός του ταμείου, οπότε θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάποιες προτιμήσεις, κάποιο πρόγραμμα, δηλαδή στείλει ένα σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα, με την γεωργία και, και οτιδήποτε είναι επιστροφές ε, θα μπορούσε να δεσμευτεί για μια συγκεκριμένη χρήση. Οπότε θα μπορούσε να αποτελέσει άρα το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη την πρώτη μας προτεραιότητα. Και έτσι οι συνάδελφοι και από τη Γεωργία και από το Διαρθρωτικό Ταμείο θα μπορούσαν να δεχτούν πως ε, ε, είναι κάτι το σημαντικό αυτό γιατί βεβαίως επηρεάζει και τους κατοίκους της Υπέθρου και θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε ίδιες συνθήκες ζωής για όλους τους κατοίκους της ε, Ευρώπης. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα. Ε, οι εκκλήσεις δεν έχουν νόημα. οι εισηγητές για όλα τα ζητήματα είναι ούτως ή άλλως ε, συμμετέχουν στη συζήτηση. Αλλά πρακτικά πρέπει να έχουμε μία πρόταση. Δεν πρέπει να περιμένουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο τώρα ε, το μπαλάκι είναι στο δικό μας γήπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Προφανώς τα θέματα αυτά είναι άκρο σημαντικά. Εξαρτόμαστε από αυτές τις τεχνολογίες και μάλιστα όλο και περισσότερο, καθημερινά. Η ασφάλεια στην πληροφορική είναι ιδιαίτερο σημαντική. Και έχουμε συνηθίσει να υιοθετούμε τη σκοπιά της έξωθεν επίθεσης, του λογισμικού, του software. Να μην ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και με το hardware όμως. σε οποιονδήποτε από τους υπολογιστέ μας θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο υλικό το οποίο να ε, ενεργοποιείται έξωθεν και να δίδονται συγκεκριμένες πληροφορίες. Σας ερωτώ λοιπόν, τις ανησυχίες αυτές τις έχετε υπόψη και αν ναι, τι θα γίνει για αυτό το σκοπό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τελευταία παρέμβαση η συνάδελφος Ουλσκοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι συγγήτρια για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης αυτή την περίοδο. Για την ώρα απλώς έχω πάρα πολλές συναντήσεις και συνομιλίες με πολλούς ενδιαφερομένους. Αυτό όμω που έχει προκύψει από τι συζητήσει που είχα και τα διάφορα σεμινάρια τα οποία παρακολούθησα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικέ προσδοκίε, πολλέ προσδοκίε από εμά, για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Μπορεί να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα τη απασχόληση, τη οικονομική ανάπτυξη, τη εσωτερική αγορά. Αυτέ οι προσδοκίε είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα υψηλέ. Όμως έχουμε συναντήσει εκπροσώπους των κρατών μελών που πιστεύουν ότι πολλά πράγματα ήδη σωστά λειτουργούν και δεν θα πρέπει να παρέμβουμε. Άρα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε τις καταλληλότερε προτάσεις, όμως δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία. Και ήθελα τα δικά σα σχόλια από αυτού, διότι ανέκαθεν ξεκινούμε με υψηλότερε προσδοκίε. έχουμε το βλέμμα μας τραμμένο προς, τον, προς τους εθέρες, αλλά τελικά δεν καταφέρνουμε να μετακινηθούμε ούτε ένα χιλιοστό. Έχετε να μας πείτε λοιπόν κάτι γενικό και ενθαρρυντικό για τα θέματα αυτά. Πρώτη τελευταία η κυρία Ουλσκοκ, γιατί η κυρία Μέρκης θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Επίτροπε. Ναι. Πάρα πολλά εθνικά κοινοβούλια όπως ε, και το Ολλανδικό εξέφρασαν ε, την απογοητευσή τους γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις προς ε, την ψηφιοποίηση και βεβαίω είναι και το δικό σας πρόγραμμα αυτό. Και θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με τι εταιρείε τηλεπικοινωνία για την διαχείριση των δεδομένων από του έξυπνου μετρητέ και τα έξυπνα δίκτυα. Λοιπόν. Επίση, το μέσο αυτό συνδέοντα στην Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα, όπω ε, το σιδηροδρομικέ γραμμέ, αλλά και τα δίκτυα μεταφορά ενέργεια. Θέλω να σα πω λοιπόν με όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία έχετε, τι γίνεται με την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ειδικά αν αυτά τα διαχειρίζονται οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Σας ευχαριστώ, κυρία Μέρκης. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Επίτροπος. Thank you. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καινούργιο όλα αυτά και είναι ένα συνέστημα που το έχω εδώ και 3,5 χρόνια, ότι ζούμε το ίδιο ταξίδι. Η επιτροπή αυτή δική σας δεν χρειάζεται καν να συζητήσει τη σημασία της ε, ψηφιακής ε, μετάβασης, ε, της διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια. Είναι αυτονόητα. Καταλαβαίνετε πόσο οριζόντιος είναι ο χαρακτήρα των θεμάτων αυτών, ότι αφορά όλους τους πολίτες και κατά τη δική μου άποψη είναι ο ιδανικός τομέας όπου μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί έχει νόημα να υπάρξει ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ψηφιακή μετάβαση. Και πραγματικά ότι υπάρχουν αλληλοσυσχετισμοί με όλους τους υπόλοιπους κλάδους και τομείς. Την ενέργεια, την υγεία, τον πολιτισμό και ούτω καθεξής. Πέραν αυτού, επειδή έχω ούτως ή την εντύπωση ότι με στηρίζατε και είμαι βεβαίως ευγνώμων γι' αυτό, πέραν αυτού είμαι τέτοιος χαρακτήρας που όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και περίπλοκα, τότε γίνομαι ακόμη πιο αγωνιστική. Θα έπρεπε βεβαίω να το θέσω διπλωματικότερα. Αλλά η ελήφθη απόφαση από το Συμβούλιο όχι να χρησιμοποιηθούν νέε ευκαιρίε, αλλά κοιτάζοντα με το βλέμμα στραμμένο προ το παρελθόν. Ευτυχώ το προσφατότερο συμβούλιο τη περασμένη εβδομάδα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ένα blueprint, όπω το έλεγα, ένα αποτύπωμα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν τι διακυβεύεται εδώ. Μιλάμε για ενιαία ψηφιακή αγορά. Βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματο. Είναι κάπως αντιφατικό όλο αυτό, όμω συνεχίζω να είμαι ευγνώμων για τη δική σα ε, στήριξη και την επικοδομητική, την δημιουργική σα ε, συνεισφορά. Όλοι έθιξαν το θέμα αυτό καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι. Πάντως, θυμάμαι ακόμη την πρώτη πρώτη μας συνάντηση, τον γύρο συναντήσεων που έχουν οργανωθεί όλα αυτά τα χρόνια με την Επιτροπή σας και θυμάμαι ότι είχα καθορίσει μια πορεία για να μπορεί κάθε Ευρωπαίος να έχει πρόσβαση την ψηφιακή τεχνολογία. Το είχα πει τότε και παραμένει γεγονός και ακόμη έχει νόημα. Δεν θέλουμε να υπάρχει κατάτμιση, δεν θέλουμε να υπάρχει κατακαιρματισμός ούτε διχασμός. Δεν θέλουμε κάποιο που ζει στην Ήπεθρο να είναι πολίτη δευτέρα κατηγορία. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί. Φανταστείτε. Το είπε ο κύριο Σέλλερ. Δίνουμε ευκαιρίε στου πολίτε και όλοι το θίξατε αυτό. Δίνουμε ευκαιρίες λοιπόν στους πολίτες. Αλλά αν τις δίνουμε, δεν πρέπει να υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση, ούτε βάση ηλικία ούτε κάτω μέλους κατοικία, ούτε περιοχής υπαίθρου ή αστικής. Και πάλι όλα αυτά σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία, με τον πολιτισμό, με την ενέργεια. Εάν υπάρξει παραμικρή διάκριση, αυτό είναι τεράστιο σφάλμα, διότι έτσι δεν δίδονται οι ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Αυτές που έχουμε υποσχεθεί, τη διασύνδεση. Να μιλήσουμε τώρα για το CEF. Είναι ένα συναρπαστικό, ένα υπέροχο εργαλείο. Γιατί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είχαμε εντατικές συζητήσεις με 9,2 δις ε, ευρώ πρόταση για την ευρυζωνικότητα. Σε αυτό θα υπήρχε και η μόχλευση με, δημιουργικό, με αυτό το δημιουργικό εργαλείο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τότε φτάναμε τα 80 δις. Και αυτό θα είχε νόημα κυρία Πρόεδρε. Αν είχαμε 80 δις ευρώ ειδικά για αυτό το θέμα, με αυτό το ποσό, τότε στις περιοχές της Υπέθρου, σε όλες τις περιοχές που κλασικά δεν αποτελούν για τις ιδιωτικέ εταιρείε στόχο προτεραιότητας, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό ήταν το πρώτο σφάλμα στη συλλογιστική του Συμβουλίου. Τα παραβλέπουν αυτά χρησιμοποιώντα το επιχείρημα ότι ε, εντάξει, ούτω ή άλλω αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δουν οι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Όχι δεν τα δαπανούν τα χρήματά τους σε μη κερδοφόρες δραστηριότητε. Μπορώ να φανταστώ και γιατί και στην περίπτωσή μας έχουμε ευθύνη. Μιλήσαμε για τα ωφέλη σε κοινωνικό επίπεδο και πώς μπορεί αυτά να είναι θετικά. Γι' αυτό είπα και εγώ για τις επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές και τους τομείς της υγείας, της ενέργειας και του πολιτισμού. Είμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Λιγότερα από 80 δις ευρώ για τις περιοχές της υπαίθρου σε αυτόν τον τομέα. Αυτό που τώρα διακυβεύεται και σωστά το είπατε κι εσείς, πήγαμε από τα 9,2 στο 1. Σαφές μήνυμα δεν κατάλαβαν τι διακυβεύεται. Αυτό μπορούμε να τους πούμε. Εγώ τίνω να έχω ενοχές κατά καιρού και διαρωτώ με μήπως δεν το εξηγήσαμε αρκετά καλά τι συζητάμε εδώ αλλά αυτό είναι πια στα χέρια μα. το Αυτή την ευθύνη πρέπει να τη δούμε και πρέπει να βρούμε μια παρακαμπτήριο για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό έχω κατά νου και γι' αυτό έκανα αυτές τις προτάσεις. Για όλους τους ενδιαφερομένους, συνάντησα συναδέλφους σας, επιτρο... Ε, προέδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών, επικεφαλής πολιτικών ομάδων, προσπάθησα να καταστήσω σαφές ότι και με τα προγράμματα τα των διευθυντικών ταμείων μπορεί να προκύψει χρηματική συμβολή εδώ, χρηματοδότηση. Και αυτή η επιλογή θα είναι ενδιαφέρουσα εφόσον η ευρυζωνικότητα και η πληροφορική με την επικοινωνία και τις ε, τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία αυτό το σύνολο λάβουν χρηματοδότηση και από τα ταμεία. Βεβαίω, το Συμβούλιο μόλι πρότεινε κάτι τέτοιο, αλλά για να το καταλάβουν και εκείνοι στη δική του γλώσσα, ελπίζω θα βοηθήσετε κι εσεί. Θα δραστηριοποιηθείτε σε αυτή την ε, κατεύθυνση, διότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, μπορείτε να πιέσετε, να προωθήσετε τέτοιου είδους διαδικασίες, ώστε να καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα. Η περίοδος αυτή είναι γεμάτη προκλήσεις. Οι προσεχείς μήνες, ιδίως το δίμηνο πριν τις διακοπές, είναι ζωτική σημασία για να δημιουργήσουμε μια ευκαιρία και να μην υπάρχει πραγματικά διχασμός στην Ευρώπη όταν μιλάμε από την σκοπιά της ψηφιακής μετάβασης. Κοιτάζω τώρα τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις σας, τις σκέψεις και τις δημιουργικές σας προτάσεις και πραγματικά το Συμβούλιο δεν φαίνεται να παραδέχεται πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά ενιαία ψηφιακή αγορά, τηλεπικοινωνίες, το οξυγόνο για, το, για την οικονομία του μέλλοντος. Αυτό εννοώ. Και την επιθυμία του Συμβουλίου την σημειώνουμε. Θα φροντίσουμε να υποβάλουμε σχετική πρόταση ως το επόμενο Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Ρώτησες, Πιλάρ, τι σκοπεύετε να κάνετε για το blueprint, το αποτύπωμα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα εδώ για τα οποία προσπαθούμε να βρούμε κάποιες πρώτες ιδέες, αλλά είναι σαφές. Όταν μιλάμε για την αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι... Μιλάμε για συλλογή 27 διακριτών εθνικών αγορών. Υπάρχει κατα... κατακαιρματισμός μπορούμε να το πούμε αυτό. Τι σημαίνει ο κατακαιρματισμός. Σημαίνει ότι είναι λιγότερες επιλογές των καταναλωτών, αλλά και για τις επιχειρήσεις, για, τους, ε, για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον εκτήματα στο να διοργανωθούν πανευρωπαϊκά. Οι χώρες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις δεξιότητες και στην ε, διακρατική ανταγωνιστικότητα. Τώρα, αυτό που μου θυμίζει όλο αυτό είναι ότι θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με τις τραπεζικές δραστηριότητες, κάτι που πρότεινε και ένας συνάδελφός μου, Τραπεζική Ένωση. Εάν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε πρόταση όπου το ίδιο είδος προσέγγισης να ακολουθείται και εδώ, θα ήταν καλό. Ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς των ψηφιακών επικοινωνιών αλλά θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι ίσως έτσι να τονωθεί η οικονομία μας κατά 210 δις ετησίως. Εάν έχει κανείς επίγνωση αυτής της ευκαιρίας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να, το, να την αδράξει. Ακολουθώντας και τις συστάσεις του Συμβουλίου, θα, θα προχωρήσουμε λοιπόν με το ανάλογο πακέτο μέτρων, τη δέσμη μέτρων, θα τα παρουσιάσουμε και σε εσά και είναι το χρόνο ώστε πριν την σύνοδο του Οκτωβρίου να δούμε, να δούμε εάν ακριβώς αυτό θέλαμε να πετύχουμε, για να πιέσουμε. Να δημιουργηθεί, να ολοκληρωθεί αυτή η αγορά. Μιλώντας τώρα για την ανάπτυξη και τα ICT, τις σχετικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν εδώ δύο βασικά επιχειρήματα. Χρειαζόμαστε απελπιστικά τις γυναίκες, τις νεαρές γυναίκες σε αυτόν τον τομέα. Τι είναι ενδιαφέρον εδώ, ήδη το αναφέρατε κι εσείς. Αυτό το κομμάτι του πληθυσμού μας το έχουμε φέρει κοντά στον τομέα αυτό. Αλλά πρέπει κανείς να ξεκινήσει νωρίς, ήδη από το δημοτικό, με ανάλογες δραστηριότητες, ώστε να είναι ξεκάθαρο. Αυτού του είδους η προσέγγιση Και είναι σαφές ότι τα κορίτσια άνω των 10 είναι πολύ έξυπνα στο χειρισμό των γκάτζετ, όπως και τα αγόρια. Αλλά για κάποιες δεν είναι αρκετά ελκυστικό να ακολουθήσουν αυτή την, την πορεία και για το μέλλον, για τη σταδιοδρομία τους. Όταν λοιπόν μιλάω για την πρωτοβουλία για τα κορίτσια στον τομέα των επικοινωνιών και της, πληροφορία, της πληροφορικής και της τεχνολογίας, Πρέπει να ξεκινήσουμε νωρί. Ξεκινήσαμε συνεργασία με τον ε, ενδιαφερόμενο κλάδο, με τα πανεπιστήμια. Ε, δημιουργήσαμε ενό είδου συμμαχία, ένα συνασπισμό, ζητώντα από τι εταιρείε με δράση στον τομέα αυτό να συγκεντρώσουν ε, τις προσπάθειές τους ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα του πώς το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Από τη μια να αντιμετωπίσουμε τους απαράδεκτους αριθμούς ε, ανεργίας τους νέους και από την άλλη γνωρίζοντας ότι ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν όταν υπάρχουν δεξιότητες ICT και τις χρειαζόμαστε να τις καλύψουμε τις θέσεις αυτές πριν το 2015. Πρέπει λοιπόν να είμαστε δραστήριοι για την πρωτοβουλία αυτή. Και στο και στην έκθεση πληροφορικής στο Ανόβερο όπου οι βουλευτές έκαναν εξαιρετική δουλειά για να παρουσιάσουν και να πούμε τι είδους θέματα πρέπει να ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτυχθούν για να έχει κανείς ένα ολοκληρωμένο CV, ολοκληρωμένο βιογραφικό Έτσι έγινε κατανοητό ότι αν κανείς ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση μπορεί να είναι και τυχερός και να βρει μια δουλειά. Όπως ε, είπε και η Σίλβια για το θέμα αυτό, και το είπα και εγώ στις εναρκτήριες παρατηρήσεις μου, Πιλάρ, ελπίζω ότι θα είναι σύντομα έτοιμη η έκθεσή σου. Είναι ζωτική σημασία να το δούμε αυτό. Χθε το βράδυ συναντήθηκα με τον πρόεδρο Τόμα Σίλβερ. Με ε, μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τον έφος. μου εξήγησαν ότι σε ένα δίμηνο περίπου θα έχουν πιο συγκεκριμένε προτάσεις. Θα παρουσιάσουν τις πρώτες προτεραιότητες στο τι πρέπει να γίνει. εξαιρετικέ ε, γνώσεις οι συμμετέχοντες στην ομάδα αυτή αλλά και ο πρόεδρος της Εστονίας ενδιαφέρθηκε πολύ για το θέμα αυτό και για την ηλεκτρονική υγεία το ίδιο, εξαιρετικά αποτελέσματα τώρα. Πρέπει να πιέσουμε λοιπόν για το νέφος τώρα, για το ηλεκτρονικό νέφος και να έχουμε πάντα υπόψη εδώ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την πλευρά του κόστους. Αυτό σχετίζεται και με την ασφάλεια στον χώρο. Θα πηδήξω εδώ λοιπόν σε ένα άλλο θέμα όπου γνωρίζουμε ότι αρκετοί Ευρωπαίοι δεν έχουν ποτέ μπει στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Ένα παράδειγμα. Έχουμε και άλλα αποτελέσματα. Στην Ιταλία μόνον το 40%, το 40 του Ιταλικού πληθυσμού δεν έχει ποτέ επισκεφτεί τον κυβερνοχώρο. Αυτό τι είναι. Μήνυμα είναι ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Οι λόγοι κάποιες φορές είναι ότι υπάρχει καχυποψία ή σκέφτονται οι άνθρωποι ότι δεν κάνει για αυτούς ή ότι δεν είναι αρκετά ασφαλές. Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, να το καταλάβουν ε, και πρώτη η Ιταλική κυβέρνηση. Ιδίω ο αρμόδιος υπουργό. Πρέπει να πιέσουμε, να υλοποιηθούν αυτά αυτά που έχουμε ως προτεραιότητα και περισσότεροι Ιταλοί πολίτες να καταλάβουν τι πλεονεκτήματα ε, μπορεί να τους δώσει η χρήση του ε, ίντερνετ. Αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όταν ε, μιλάμε για την στρατηγική που καταρτήσαμε από κοινού με τη Λέδη Άστον και την Σεσίλια Μάλστρομ ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελπίζουμε ότι εδώ πάλι με την συμβολή του Κοινοβουλίου θα καταστήσουμε σαφές ότι αυτή η προτεραιότητα πρέπει να ε, προχωρήσει. Mrs. Um, was for Η κυρία Καρβάλιο μίλησε στην ανοιχτή πρόσβαση, στην ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσίευσεις. Έχουμε κάνει καλή δουλειά μιλώντας ε, για την ελεύθερη πρόσβαση σε επιστήμονες. Θα θέλαμε να υπάρξει μεγαλύτερη ε, πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση για τους περισσότερους, να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται να υποβάλουμε πρόταση για το κόστος σχετικά με το θέμα αυτό και ένα πολύ σύντομο σχόλιο ότι όλοι εκνευριζόμαστε όταν ε, γίνονται έργα σε ένα δρόμο για να ε, γίνουν ε, επισκευές στο σύστημα ενέργειας, αλλά μετά από μια εβδομάδα είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κερδίσουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με ένα καλύτερο συντονισμό στα έργα και τις επενδύσεις. Έτσι μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση των επενδύσεων και αυτό θα καλυφθεί και στις υπόλοιπες πρωτοβουλίε μας του Οκτωβρίου. Το έχουμε στον κατάλογό μας. Το Horizon 2020 θα επικεντρωθούμε προφανώς στην ελεύθερη και ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση. Ο κύριος Πρόντι ανέφερε το τι γίνεται με το hardware και πώς σχετίζεται το θέμα αυτό με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αποτελεί βασική προτεραιότητα στον κατάλογό μας. Εάν δεν υπάρξει ασφάλεια, δεν θα υπάρξει και πρόοδος. Πολλοί, όχι μόνο στην Ευρώπη και εκτός, ενδιαφέρονται, καραδοκούν να βρουν τις αδυναμίες μας, να εντοπίσουν αδυναμίες στο σύστημά μας. Υπάρχει λοιπόν Ε, ε, παγκόσμιο ενδιαφέρον σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο για την ασφάλεια στην, στον κυβερνοχώρο. Διαφέρει από το έγκλημα το κλασικό, το συνηθισμένο, η επίθεση, η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες λύσεις εύστοχες το ίδιο και με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Θέλουμε να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Θα χρησιμοποιούνται περισσότερο ψηφιακές υπηρεσίες εάν βελτιωθεί η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αυτό θα ενισχύσει και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητά μας και την ενοποίηση της ε, ψηφιακής αγοράς. Επίσης, θίξατε το θέμα το θέμα των ευθειών πόλεων και το πώς μπορούμε και τις τεχνολογίες και τις μεταφορές και την κινητικότητα και την τεχνολογία να τα συνδυάσουμε. Για να συμβάλλουμε στους στόχους του 2020 στην ενέργεια. Οπότε, γι' αυτό και επιμένουμε σε κάποιες λύσεις σε σχέση με τα προαπαιτούμενα για μια διαλειτουργικότητα, ώστε να μπορούν να συνομιλήσουν, να συνεργαστούν οι πόλεις και όσον αφορά τις υποδομές για όλους τους χρήστες και όπως θα πρέπει να υπαρρυπνεί πάσα πόλη για τις αριστερές ε, πρακτικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας που νομίζω ότι κάλεψαν όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα εργαστούμε τους προσεχείς μήνες μαζί μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι και το ίδιο και οι συνάδελφοι. Bene, con i nostri lavori. Ωραία. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Το λόγο έχει η κυρία Ουλσκοκ, η οποία θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Ντόχα, τη συμμετοχή δηλαδή, το Δεκέμβριο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω τι έγινε. Τρεις πριν τρεις μήνες πήγαμε στην Τόχα. Και το θέμα βέβαια είναι να προετοιμαστούμε για την επερχόμενη συνεδρίαση. 15 πήγαμε στην Τόχα. Ε, μέλη της Επιτροπής. Ήτρα είχαν πολύ εντατικό πρόγραμμα, έξι μέρες στην Τόχα. Συναντήσαμε τον Επίτροπο. Την Κυπριακή Προεδρία, την Ιρλανδική Προεδρία και άλλους εκπροσώπους του Συμβουλίου βεβαίως. Βεβαίως, ε, ε, είδαμε την ηγεσία του Κατάρ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Βραζιλίας και εκπροσώπους και άλλων χωρών. Ο δε Κινέζος Υπουργός μας είπε πως οι Κινέζοι πιθανώς να σκεφτούν ε, να ενταχθούν σε ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών που θα μπορούσε ακόμα και να συμπεριλαμβάνει και την αεροπορία. Φοβέρες καινοτομίες. Και τώρα βεβαίως θα πρέπει η Επιτροπή Περιβάλλοντος να δει αν ε, πηγαίνουν πουθενά όλες αυτές οι υποσχέσεις. Ήταν ε, αποτελεσματικό λοιπόν το έργο μας, θα έλεγα, ως ε, επαφές είχαμε και τις δικές μας επαφές, ένα σεμινάριο για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο των δύο βαθμών θερμοκρασίας. Επίσης, συναντήσαμε πάρα πολλές ΜΚΙΟ και είχαμε σειρά εργαστηρίων όπου συνομιλήσαμε με προσώπους της βιομηχανίας, Τι έγινε λοιπόν στην ε, συνάντηση αυτήν. Ήταν απογοητευτική. Αλλά ε, όσοι έχουμε πάει σε αρκετέ τέτοιε συναντήσει δεν απογοητευτήκαμε τόσο γιατί παρόλα αυτά ήταν σαφές πως η συμφωνία του Κιώτο που δεν ε, έχει απομείνει πλέον με πολλά κράτη-μέλη αλλά είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία παρατάθηκε έτσι περαιτέρω, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Οπότε το ζήτημα τώρα είναι τι κάνουμε με τα λοιπά δικαιώματα εκπομπών της πρώτης περίοδου του Κιώτο και θα είναι πιο δύσκολο να τα εμπορευθούμε αυτά αλλά επιτευχθεί ακόμα και εκεί πέρα πρόοδος υπήρξε ένα αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πρόγραμμα εργασίας για φέτος, για να μπορέσουμε κάποτε να συμφωνήσουμε σε μία πρόταση που θα ολοκληρωθεί το 2015. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς λόγω της συνόδου που θα λάβει χώρα στην Ευρώπη. Και εκεί πέρα θα ληφθούν η αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούμε το σύστημα και το τι θα γίνει για να έχουμε μια συμφωνία την οποία θα μπορέσει να υποστηρίξει και ο κόσμος. Η επόμενη σύνοδος λοιπόν θα είναι το Νοέμβριο στην Βαρσοβία, στην Πολωνία, επί ευρωπαϊκού εδάφους θα έχουμε ηγέτες από όλο τον κόσμο. Και βεβαίως ε, θα έχουμε και μια συνάντηση που θα φιλοξενήσει η ε, Γαλλία. Δεν υπάρχει λοιπόν πάρα πολύς ε, χρόνος και δεν ξέρουμε το τι θα κάνουμε για να ανταποκριθούμε και στις δικές μας τις δεσμεύσεις που εδώ και πολύ καιρό έχουμε αναλάβει. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτές τις συναντήσεις σωστά. Δεν είχαμε τίποτα φοβερά νέα, αλλά συνεχίσαμε να πιέζουμε, έγιναν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπήρχαν και άλλα ζητήματα και ε, δεν ε, εμφανίστηκαν όλα αυτά στα μέσα, αλλά νομίζω πως ε, τώρα βεβαίως στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας. Το 2013 είναι η πρώτη στιγμή, αν θέλετε, Τη αλήθεια. 2014 από τη Σύνοδο Κορυφή με αρχηγού κατών και κυβερνήσεων τον Μπαν Κιμούν άλλη μια αποφασιστική στιγμή και τέλο το 2015 που θα φιλοξενήσει η Γαλλία την ε, σχετική σύνοδο έχουμε άλλη μια σημαντική ημερομηνία και πρέπει να έχουμε μια συμφωνία ε, όπως είπα ε, που θα τύχει ευρεία στήριξης θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Ρίντσε, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ με τη δική του έκθεση. Και τώρα το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε τους επόμενους 8-9 μήνες, έτσι ώστε εμείς ως Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα βήματα για να προχωρήσουμε προς την Βαρσοβία. Να δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να έχουμε άλλο ένα δίκτυο στις επιτροπές περιβάλλοντος και λοιπόν για να δούμε το τι θα γίνει. Ε, άνθρωποι οι οποίοι όχι οπωσδήποτε θα ταξιδεύουν αλλά θα εργαστούν επί του θέματος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο και να καταλήξουμε τότε σε ψήφισμα που θα αποτελέσει την εντολή του Κοινοβουλίου πρέπει να ξεκινήσουμε από νωρίς. Και ελπίζω όλοι μας να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς ένα σχέδιο το οποίο θα μας επιτρέψει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε λίγα λεπτάκια, όχι πάρα πολλά γιατί όπου να είναι θα έρθει ο κύριος Έτιγκερ Λοιπόν, η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έλαβα μέρο σε αυτήν την προσωπία. Ακριβώς όπως έλεγα. Τα βασικά συμπεράσματα ήταν η δεύτερη περίοδο δέσμευση για το πρωτοκόλλο του Κιώτο και επίση είχαμε και κάποιε άλλε αποφάσει όσον αφορά τη χρηματοδότηση και αυτό βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά τα όσα ανακοίνωσε ε, η Αγγλία και η Γερμανία όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αναπτυσσομένων χωρών και τώρα όσον αφορά την πλατφόρμα για την ανάπτυξη. Αυτά δηλαδή που θα γίνουν την επαύριο της περίοδου του Κιώτο δεν είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο κυρίω όσον αφορά ε, το χρονοδιάγραμμα, τα διαδικαστικά, τα μεθοδολογικά και πρόκειται ακριβώ για το ότι ακόμη, ακόμη η κατάσταση είναι θολή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την πλατφόρμα για την ανάπτυξη. Είναι ευκαιρία πάντω όλα αυτά για την Ευρώπη, ούτω ώστε να μπορέσει, να μπορέσει να έχει την, ε, να μπορέσει να έχει την πρωτοβουλία στι εξελίξει, το πρωτόκολλο του Κιώτο. Εστέζει κυρίω όσον αφορά τα κλιματικά. Θα πρέπει όμως να λεφθούν υπόψη και τα θέματα τη ανταγωνιστικότητα. Άρα ας προετοιμαστούμε να καλύψουμε και ένα τέτοιο μοντέλο που θα αφορά την ανταγωνιστικότητα σε οικονομία, σε βιομηχανία, σε, σε εξασφάλιση των προμηθειών. Άρα θα πρέπει η Επιτροπή να ετοιμαστεί γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία τώρα αντιγυμνοζήμασουν για την οικονομία της Ευρώπης. Stiamo al massimo i due Παρακαλώ δύο λεπτά για ε, να μην περιμένει ο Επίτροπος. Έχετε το λόγο κύριε. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε σωστή παρουσίαση της κατάστασης, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Ε, στο Κοινοβούλιο έρχονται πάντα τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στο τέλος του έτους υπό μορφή ψηφίσματος. Πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε από τώρα και εδώ πέρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω κυρία Πρόεδρε να γίνει η προετοιμασία του ψηφίσματος στην Επιτροπή μας παράλληλα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί υπάρχουν πάντα εντάσεις. Τώρα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε πώς θέλουμε να έχουμε έναν ισότιμο ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βεβαίω θα δούμε και τις διάφορες αρμοδιότητες που υπάρχουν και θα δούμε τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Ο κύριος Έλμερ, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία και όχι κυρία. Φαίνεται, ότι ξεχάσαμε την πραγματικότητα έξω στον πραγματικό κόσμο και η πραγματικότητα είναι ότι παντού σε όλο τον κόσμο έχουμε 1200 τέτοι, τέτοιους σταθμούς οι τώρα κατασκευάζονται και θα βασίζονται στον άνθρακα. Και έχουμε όλες αυτές τις διασκέψεις στις οποίες πάμε και ερχόμαστε και εκεί πέρα έχουμε αυτούς τους ε, ειδικού οι οποίοι τα λένε μεταξύ τους και αγνοούν την πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα στον κόσμο κανείς δεν, δεν πιστεύει σε αυτά που λένε, κανείς δεν τους ακούει. Και, έχουμε τον δόκτορα Τσα, Τσαπάρη της IPCC ε, και μας λέει εδώ και 17 χρόνια για την υπερθέμιση του πλανήτη και όλα αυτά. Μα καλά, πόσο, πόσο και θα το πηγαίνουμε έτσι το πράγμα. Και αν είχαμε βέβαια κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, ε, μειώσεις του διοξιδίου του άνθρακα, τότε θα έπρεπε να, να, να περικόψουμε και όλες τις εκπομπές της λαπτικές, τις 20.000 πόσο είναι τόνους, ε, που εκπέμπουν πηγαίνοντα στο Στρασβούργο. Και επομένω αυτό θα πρέπει να γίνεται και να σταματήσουμε αυτά τα ταξιδάκια σε εκδρομέ, σε αυτέ τι διασκέψει πάντω στον κόσμο. Ευχαριστώ. Πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλουμε να αναθεωρήσουμε 100% την άποψή μας, διότι το πρωτόκολλο του Κιώτο επίσημα ισχύει, αλλά όλο ένα και λιγότερες χώρες το υλοποιούν. Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μια γενική διαπίστωση μια από το πρωτόκολλο του Κιώτο δεν λαμβάνει υπόψη την διακήρυξη του Μπαλί για την συνυπευθυνότητα. Άρα, να ξαναρχίσει η ζήμωση, λαμβάνοντα και αυτό που σα είπα υπόψη. Έτσι μόνο θα φτάσουμε σε μια παγκόσμια συμφωνία, γιατί χωρί παγκόσμια συμφωνία θα πρέπει να βρούμε το plan B, το εναλλακτικό σενάριο. Θα πρέπει επομένω αυτού του είδου η συμφωνία παγκόσμια να είναι το σενάριο Α. Αν όμω δεν πετύχει κάτι να έχουμε ένα πλάν B εναλλακτικό. Αλλά θα πρέπει, οτιδήποτε, για το πλάνο Α θα πρέπει να υλοποιήσει, να γίνει πολιτική πράξη το πρωτόκολλο, η απόφαση του πάντων του Μπαλί. Ο επόμενο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέει ο κύριο Οντή, Άκουσα ότι είπε η κυρία Καρβάλιο ότι θα πρέπει όντω να διαρθρώσουμε ε, να περιστρέφεται τέλο πάντων η πολιτική ζήμωση γύρω από όλα αυτά, γιατί ψηφίζουμε για αυτή μας την έκθεση για τι ανανεώσιμε πηγέ, ενέργειες, τα αυτοκίνητα και στι μας μα. Ε, Δυσκολεύομαστε πάρα πολύ να βρούμε μια ρότα και η πολιτική μας γραμμή ακόμα δεν έχει εξευρεθεί. και τέλος του 2008 ας πούμε εγκαταλείφθηκε τότε η πολιτική γραμμή από τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων όσον αφορά ε, το τι θα γίνει με τα περιβαλλοντικά. Τώρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε ενώ στην εκλογών του 2014 να δούμε τι, τι, τι προβληματική θα γίνει και έτσι να ετοιμαστούν οι επόμενες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το επόμενο κοινοβούλιο. Θα πρέπει επομένως ακόμα να κάτσουμε να βρούμε όλους τους άξονες που θα περιστρέφει μας μας πολιτική για ανάπτυξη, για ανταγωνιστικότητα, για όλα αυτά που έχει να εντοπίσει την παγκοσμία σκηνή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι να διαρθρώσουν την, την, πολιτικό, την πολιτική μαζί μας. Και τώρα επομένως, ας καλωσορίσουμε τον ε, Επιτροπό Έντιγκερ και θα μας μιλήσει μας κάνει την εισήγησή του. Κύριος Οέτιγκερ. Bene, diamo allora... Ωραία. εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής, τον Επίτροπο Έτιγκερ επιφορτισμένο με θέματα ενέργειας. Θα μας μιλήσει εδώ για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και το τι θα κάνουμε μαζί. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, έχετε 15 περίπου λεπτά για την εισηγήσή σας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι ε, δεχτήκατε την πρότασή μας ε, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα προστασίας ε, του περιβάλλοντος. Γνωρίζοντας πως πρέπει να ε, έχουμε και ασφάλεια και στην παραγωγή πετρελαίου στα δικά μας χωρικά ύδατα, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα. Και άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για την πρόληψη και για την έκτακτη περίπτωση. Οπότε έχουμε άλλο ένα βήμα περαιτέρω στον εξευρωπαϊσμό της πολιτικής ενέργειας και περιβάλλοντος. Και θα με ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήταν εδώ πέρα αρμόδιοι. Πού είναι το βάρος που δίνουμε λοιπόν στις εργασίες μας φέτος. θέλουμε το ενδιαφέρον να μετατοπιστεί από το 2020 στο 2030. Όποτε μιλάω με πολιτικούς που ασχολούνται με την ενέργεια και με τον κλάδο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη ασφάλεια σχεδιασμού. Εξακολουθούμε βεβαίως να ελέγχουμε την τήρηση των στόχων του 2020 και υποβάλλονται και τακτικές εκθέσεις προόδου. Αλλά τώρα έχει φτάσει η στιγμή να γίνει η συζήτηση για μια ευρωπαϊκή ε, στρατηγική ενέργειας και κλίματος πέρα από το 2020. Γιατί το εξή είναι σαφές. Εάν δεν υπάρξει μια τέτοια στρατηγική, τότε η όλη υπόθεση κοινή ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής έχει τελειώσει. Θα καταλήξουμε σε κατακαιρματισμένες αγορές, διαφορετικές εξελίξεις στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τελικά δεν θα κάνουμε τίποτα όσον αφορά την μείωση κομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ξέρετε πως... Ε, την Τετάρτη που μας έρχεται, σε μία βδομάδα, θα έχουμε την υποβολή μιας πράσινης βίβλου από την Κομισιόν, από εμένα και την κυρία Χέντεγκαρντ. Ορίζουμε κάποιους στόχους και κάποια ερωτήματα και απευθυνόμαστε και προς εσάς, προς το Κοινοβούλιο. Και θέλουμε, με βάση τις διάφορες συνθέσεις που υπάρχουν. Π.χ. Ε, μετά το Πάσχα έχουμε άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, έχουμε κοινή συνεδρίαση Συμβουλίου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θέλουμε εκεί στο Συμβούλιο να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις που θα γίνουν νομοθετικές προτάσεις προς το τέλος του έτους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα στόχο για τις εκπομπές και ένα στόχο για τις ανανεώσιμες και έναν στόχο για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Η πράσινη βίβλος ε, θεωρεί πως υπάρχουν κοινοί στόχοι, δηλαδή ασφάλεια στην ε, προμήθεια, αηφορία και προσιτές τιμές για ρεύμα και φυσικό αέριο. Νομίζω πως ε, Ε, δεν θα πει κανεί, δεν θα έχει κανεί να προχωρήσουμε σε ένα πολύ πιο φιλόδοξο στόχο για μετά το 2020, ε, για μείωση των εκπομπών. Τώρα, για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Χρειαζόμαστε υψηλότερο στόχο. Εγώ είμαι ανοιχτό. Αλλά θεωρώ πω η ενεργειακή μα πολιτική δεν πρέπει να είναι μόνο μείωση των εκπομπών. Όσο σημαντική και αν είναι αυτή, πρέπει να προωθήσουμε και τι νέε τεχνολογίε και την καινοτομία. Και Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση με τις ε, ανανέσιμες πηγές ενέργειας. Οπωσδήποτε ηλιακή, αιωλική, οπωσδήποτε η ενέργεια των κυμάτων, ε, τα υδροηλεκτρικά, η γεωθερμία, ειδικά τα τελευταία που ανέφερα πρέπει να εφαρμοστούν, ειδικά στη Γαλλία, ξέρετε και η Ιρλανδία, η ενέργεια των κυμάτων ε, ήδη ε, αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης. Το ζήτημα είναι λοιπόν τι στόχος θα πρέπει να είναι ο στόχος των ανανεώσιμων. Ένας στόχος παραγωγής ρεύματος, ένας στόχος των μεταφορών, ε, σε ποιο πεδίο. Εδώ πέρα αναμένω την δική σας την συνεισφορά και γενικώ αυτό το οποίο με ενισχύει περισσότερο είναι το εξής. Το 2007 όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν. Πώς θα έχουμε σε 28 κράτη-μέλη μια κοινή ε, πολιτική και θα συμφωνήσει και μια ευρεία πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάναμε Ε, θα κάνουμε συγχωρείτε στο τέλος του έτους την πρότασή μας ε, στο τέλος του έτους, οπότε θα απασχολήσει κατά βάση το επόμενο κοινοβούλιο από το 2014 και μετά. Και άρα το 2015 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα το 2030. Νομίζω λοιπόν πως αυτό είναι το πολιτικά πιο συναρπαστικό θέμα για την ε, πολιτική μας της ενέργειας. Βεβαίως, για μένα το κλίμα και η ενέργεια είναι ε, ισότιμα. Αλλά ο τομέας της ενέργειας δεν υπηρετεί τον τομέα του κλίματος, αλλά είναι κάτι το ξεχωριστό και με πτυχές κοινωνικές, όπως είπα, της προσιτής τιμής, αλλά και όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την παγκόσμια διάσταση. Θέλουμε λοιπόν την ολοκλήρωση επίσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας που θέλουμε να αποτελέσει έναν δεύτερο στόχο μας και θεωρούμε πως ο σχεδιασμός της αγοράς και το ποιες εθνικές παρεμβάσεις επιτρέπουμε στο πλαίσιο των κανόνων της εσωτερικής αγοράς μέσω κατευθυντήρων γραμμών της Κομισιόν, το τι συμφωνεί δηλαδή με το δίκαιο του ανταγωνισμού και το τι ε, όχι, είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας καθοδηγούν. Δηλαδή, σχεδιασμός αγοράς, μηχανισμοί ε, για τις ε, δυνατότητες παραγωγής. Οπότε ο σχεδιασμός της αγοράς είναι μια απόκληση από την καθαρή λογική της αγοράς. Δηλαδή η εσωτερική αγορά σημαίνει προσφορά, ζήτηση, διαφάνεια και ή δυνατόν καμία παρέμβαση του κράτους, ε, δήμων κτλ. Καμία έμεση ή άμεση οικονομική ενίσχυση. Καμία προτίμηση ή ε, ε, εύνοια σε κάποια μορφή ενέργειες. Αλλά ξέρουμε πως σε μια καθαρή τέτοια αγορά δεν υπάρχουν επενδύσεις. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά υπάρχει, όπως είπα, και το ζήτημα οικοδομιστών δυνατοτήτων, ειδικά όσον αφορά το φυσικό αέριο ή το Ηνωμένο Βασίλειο πηγαίνει σε μια κατεύθυνση νέων πυρηνικών ε, εργοστασίων, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τις ε, εγγυημένε ε, τιμές για παροχή ενέργειας προς το δίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν όπως σας είπα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και θέλουμε μια εντονότερη σύγκληση των εθνικών συστημάτων προώθησης των ανανεώσιμων. Θεωρούμε πως είχαμε κάποιες καλές εμπειρίες στον τομέα αυτών και κάποιες κακές εμπειρίες που μπορούμε να μοιραστούμε. Το θέμα δεν είναι, όπως είπα, η προσέγγιση μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για κάποιες κοινέ εμπειρίες οι οποίες ε, θα, αποτελούσαν, ε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ε, υπόδειγμα, αν θέλετε, για άλλες χώρες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τις τελευταίες εβδομάδες έλαβα πάρα, πολλές, ε, πάρα πολύ επικριτική για το ζήτημα της αλλαγής των τιμών στην Ισπανία. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες εγγυημένε τιμές, κάποιοι επένδυσαν, άρχισαν να παράγουν ρεύμα και έχαναν λεφτά τελικά. Μιλάμε για απόλυες 29 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες. Οπότε η επιδότηση της ε, ηλιακής ε, ενέργειας μειώθηκε και όχι για το μέλλον, για να σχεδιάσει κανείς, για τα υφιστάμενα ηλιακά. Έτσι οι ε, επενδυτές βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση. Υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες ε, κάνουν και αναδρομικές μειώσεις. Αυτό το οποίο προτείνεται παραδείγματος χάρη στη Γερμανία. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό, το βρίσκω τελείως λάθος. Και τίστε και ζήτημα συνταγματικότητας και ιδιοκτησίας, να μην μιλήσω για την εμπιστοσύνη του επενδυτή. Εάν ισχύει κάτι και περικοπεί κιόλα αναδρομικά, τι να κάνει ο επενδυτής, τι να εμπιστευτούν οι τράπεζες, και βλάπτεται έτσι η εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρά το ότι ο κλάδος χρειάζεται περισσότερους και όχι λιγότερους επενδυτές για παραγωγή, για αποθήκευση, για αποτελεσματικότητα, για τις υποδομές. Οπότε, στο δεύτερο τρίμηνο θα υποβάλουμε την, ε, την ανακοίνωσή μας, την ερευνητική για το θέμα αυτό και θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των έργων των τελευταίων ετών από το σχέδιο Συνδέοντα την Ευρώπη μέχρι το ΙΤΕΡ και τα 7 χρόνια για τον ορίζοντα 2020. Και τελευταίο, έχω πολλά να πω αλλά θα κλείσω για την ώρα. Μετά από τα τεστ κοπόσεως των πυρηνικών εργοστασίων τον Μάιο θα υποβάλουμε μία πρόταση για την ε, αναδιατύπωση της οδηγίας πυρηνικής ασφάλειας, για προδιαγραφές ασφαλείας, με προτάσεις για μια εκτεταμένη ανεξαρτησία των ε, εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και θα καταθέσουμε και προτάσεις για την υποχρέωση ασφάλισης, για πιθανές ε, βλάβες που μπορεί να προκληθούν από βλάβες στα πυρηνικά εργοστάσια και θα δούμε ε, επίσης και τις διαφορετικές ρυθμίσεις ε, υποχρεωτικής ασφάλισης και της αστικής ευθύνης των πυρηνικών εργοστασίων στις διάφορες χώρες και Ποιε δυνατότητε υπάρχουν για τέτοιες, τέτοια, τέτοιες ασφαλιστικές συμβάσεις. Γιατί και αυτό, δηλαδή η υποχρέωση ανάληψης ευθύνης, νομίζω ε, εξυπηρετεί τον ε, δίκαιο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Αυτά λοιπόν έτσι ως ε, θέματα τα οποία είναι ανοιχτά στο πρόγραμμά μας και θα έλεγα πως ε, είστε ενημερωμένοι όχι μόνο για τα σημερινά αλλά και για τον ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας ε, και αναμένουμε βεβαίως και την πολιτική ε, συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Όπως μπορείτε να φανταστείτε έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Για να μπορέσουν όμως όλοι να μιλήσουν θα πρέπει να σεβαστείτε τα χρονικά όρια. Εάν γίνει αυτό και όλοι θα μιλήσουν και θα απαντήσει ο Επίτροπος. Για τρία λοιπόν λεπτά η κυρία Ντέλ Καστίγιο για το ΕΛΚ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε που ξαναήρθατε εδώ στην Επιτροπή αυτή, την δική σα Επιτροπή. Και Νομίζω ότι αρχίσατε κάτι να λέτε το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ότι δηλαδή η ενεργητική πολιτική είναι ενεργητική πολιτική, δεν είναι πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Άλλο το πόσο συμβάλλει η ενεργειακή πολιτική για τη μείωση των κουμπών Βέβαια είναι σημαντικό και οπότε θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η πολιτική της κλιματικής αλλαγής και το έχουμε πει επανειλημμένα και αυτό θα πρέπει να σα το πω ειλικρινά γιατί το πιστεύω ότι πρόκειται εδώ πέρα για κάποιο είδου ομοιρία υπό την οποία τελεί η ενεργειακή πολιτική ή υπό τι άλλε πολιτικέ τη κλιματική αλλαγή και ο μόνο τρόπο επομένω ε, το μόνο που χρειάζεται το μόνο για να πηγαίνει θετικά τέτοια πολιτική είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και να έχουμε λιγότερε εκπομπέ όπου και να χρειάζεται επομένω να υπάρχει τέτοια συμβολή τη ενεργειακή πολιτική ούτω ώστε να μπορεί και να συμβάλλει στην ε, αυτονομία, στην αυτάρκεια, στι υποδομέ, στο πώ θα αναπτύξουμε νέε ενεργειακέ πηγέ και επομένω έτσι να έχουμε και κάποιο είδου καινοτομία και τεχνολογία και με αυτή την ενία θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο το να. Από αυτή τη βάση να συνοηθούμε δηλαδή. Γιατί τώρα ο καθένα λέει άλλα. Και τώρα, όταν μιλούν για κοινωνική πολιτική, πώ είναι δυνατόν να μείνει κοινωνική πολιτική, ενεργική πολιτική, άμα δεν ε, ανάβει το φω, άμα δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο, γιατί δεν έχει αρκετή ενέργεια, γιατί δεν έχει τη σωστή ενέργεια, ή άμα δεν λειτουργούν οι μεταφορέ, ε, τότε είναι τρομερές, απερίγραπτες οι κοινωνικές συνέπειες. Αν δεν υπάρχει όμω μια πολίτικα τέτοια που να έχει θετικές ε, επιπτώσεις στην οικονομία και στην ε, κοινωνία, άρα και στην ανάπτυξη, ε, αυτή είναι και κατεξοχήν η ενεργειακή πολιτική. Ε, γι' αυτό σα λέω, Επίτροπε, ακόμα μένει λίγος χρόνος για αυτή τη θητεία. Οπότε θα πρέπει μέχρι το καλοκαίρι κάτι να έχει γίνει. Λαμβάνοντα υπόψη αυτήν την κατάσταση που προσφέρει να περνάμε. Θα πρέπει μόνος να χαράξουμε πορεία κατά αυτόν τον τρόπο. Για μια τέτοια ενεργειακή πολιτική. Να μην συναρτάται από άλλη, να μην εξαρτάται από άλλη. Τι προτείνει η Επιτροπή. Έτσι συμφετικά. Μας είπατε για την Πράσινη Βίβλο για, για τη συνέχεια που θα λάβει η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Έτσι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τις προτάσεις που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το, το, αργότερο θα πρέπει να έχουμε και νομοθετικές προτάσεις ε, μέχρι το φθινόπωρο. Πίλα, σε ευχαριστούμε. Τερέζα Μαντουρέλη, για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρώτα-πρώτα ευχαριστούμε που ήρθατε να μας δείτε. περισμένη εβδομάδα στο Στασβούργο ψηφίσαμε τις κινητήρες γραμμές για τις ε, υποδομές ενέργειας και είχαμε την έκθεση Κορέα Κάμπος σε σχέση με τις προτάσεις μας προς το Συμβούλιο. Πολύ σημαντική υπόθεση όσον αφορά την νέα υποδομή που θα πρέπει να υπάρχει για την ενέργεια και επίσης για το τι θα γίνει με τα προγράμματα και έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και να δούμε τι είναι τελικά επιλέξιμο για χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού συνδέω με την Ευρώπη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτέ τι ενεργειακέ υποδομέ να μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτή η πρόταση με τον Συμβουλίο και βέβαια το Συμβούλιο τώρα θέλει να περικόψει τη μισή πρικοδότηση, όμως ε, έτσι δεν υπάρχουν τα χρήματα για όλα αυτά τα προγράμματα, τα έργα που παρατηρούνται κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και γι' αυτό και η πολιτική μας ομάδα αντίθεται στο Συμβούλιο. Το επιχείρημα το οποίο λέει ότι στον ε, κανονισμό για τις συνεργειακές υποδομές ε, θέλει να αφήσει απ' έξω τέλος πάντων το Connecting Europe και να δούμε επομένω τι θα παραμείνει επιλέξιμο. Άρα θα πρέπει να έχουμε ένα άλλο μηχανισμό εκτός από τον υπάρχοντα για τις ε, δημόσιες επενδύσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό το, το έχετε και εσείς επισημάνει και ότι θα κάνει ό,τι ενέργεια χρειάζεται η, Επιτροπή για να διευκολύνει τις επαφές μας με το Συμβούλιο. Τώρα έχω άλλη μία παρατήρηση όσον αφορά ε, το, το, τη δέσμη μέτρων για ενέργεια 2030 ε, και σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρια εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας γιατί αυτό το οποίο τώρα γίνεται είναι ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες και θα πρέπει να είναι δεσμευτικά τόσο προβλέπονται. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε τυχαίο το ότι οι τρεις δείκτες, τα τρία κριτήρια για το 2020 το μόνο το οποίο θα ισχύσει τελικά είναι η προϋπόθεση, το κριτήριο, ο δείκτης που δεν είναι δεσμευτικός. Εμείς οπωσδήποτε και εμείς θα υπέρ των ε, στόχων που έχουν τεθεί, αλλά θέλουμε να είναι δεσμευτικοί. Όπως τα λέει η Επίτροπος ε, για την κλιματική αλλαγή, θέλουμε να δοκιμήσουν όσα λέει και δεν θέλουμε μια ε, πολιτική να είναι να είναι όμοιρος της άλλης και θέλουμε να είναι πραγματικά οι πολιτικές μας αποτελεσματικές. Ευχαριστούμε Τερέζα. Ο κύριος Τούρμες για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Δικαίω αναφερθήκατε στο θέμα της προσιτής τιμής της ενέργειας. Εάν δούμε τι γίνεται, βλέπουμε πως οι τιμές ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου από το 2000 ε, αυξήθηκαν περισσότερο από τις τιμές του ρεύματος ανά κιλοβατόρα. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να δούμε, αν δούμε τα νοικοκυριά, τα περισσότερα νοικοκυριά έδωσαν περισσότερα για μεταφορές και θέρμανση, δηλαδή πετρέλαιο ή αέριο, και θεωρώ πως στη συζήτηση αυτή πως πρέπει να γίνει μια κανονική ανάλυση. Εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ως Ευρώπη την παγκόσμια αγορά για το αέριο μπορούμε να ονειρευόμαστε το ότι θα εξορίξουμε τα σχιστολιθικά αποθέματα και βεβαίως ε, στο ρεύμα βρισκόμαστε σε μια φάση επανεπενδύσεων. Οπότε ακριβώς σε καιρούς κρίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Γιατί Εκεί πέρα μπορεί να μειωθεί το κόστος γρήγορα, σχετικά, και αυτό το οποίο πραγματικά μου προξενεί εντύπωση, μιλάμε για την Ευρωζώνη ή την Ευρώπη και τις αδυναμίες της. Αλλά κανείς δεν λέει για το ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε 4% του ΑΕΠ για να αγοράσουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ε, το 2000 δίναμε 1%. Δηλαδή πέφτει η ζήτηση στην Ευρώπη αλλά ανεβαίνει στην παγκόσμια αγορά. Μιλάμε για 400 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε ετησίω ε, για πετρέλαιο και αέριο και ουράνιο. Μεγάλη δυναμία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε σύγκριση με αυτό το εμπορικό μας έλλειμμα με την Κίνα είναι 120 δισεκατομμύρια. Μιλάμε κάθε μέρα για την ανταγωνιστικότητα, 120 δισεκατομμύρια δηλαδή και δίνουμε 400 δισεκατομμύρια για ε, εμπορικό έλλειμμα για την εισαγωγή ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Ε, τέλος για του ίσου ανταγωνισμού που αναφέρατε. Σήμερα δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού γιατί είναι τόσο χαμηλή η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα και για τα ηλιακά υπάρχει 100% ασφάλιση ε, και πλήρης μεικτή ασφάλιση, αλλά όχι για τα πυρηνικά εργοστάσια. Η ε, Φουκουσίμα από ό,τι φαίνεται θα κοστίσει χίλια δισεκατομμύρια ευρώ από ό,τι φαίνεται σε ζημιές. Οπότε, αν στο μέλλον τουλάχιστον στις νέες επενδύσεις θέλουμε ίσους όρου ανταγωνισμού, πρέπει να δούμε και την αστική ευθύνη των νέων πυρηνικών εργοστασίων. Και και για την πρόταση της ε, Κομισιόν μιλήσατε για την εγγύηση για τους άμεσα πληττόμενους από ένα ατύχημα. μιλάτε για τους άμεσα πληττόμενους ή για την αστική ευθύνη τη γενικότερη. Είναι τεράστια η διαφορά, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τις αποζημιώσεις των άμεσων θυμάτων μιας πυρηνικής, πιθανής ε, πυρηνικής καταστροφής. Σας ευχαριστώ κύριε Τσίτσεστερ για τρία λεπτά. Thank you, Madam ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, Επίτροπε. Χαιρόμαστε να σα βλέπουμε εδώ. Όταν η Επιτροπή αυτή είχε εγκρίνει τροπολογίε, ζητώντα από την Επιτροπή να λάβει θετικά βήματα για να προωθήσει την πυρηνική ενέργεια, παρά τι αρνητικέ απόψει του κυρίου Τούρμε για το θέμα αυτό, είναι δική μου, δικό μου χρόνο ομιλία, αγαπητέ μου, δικό μου. Τι βήματα θα λάβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακολουθήσει αυτή την τροπολογία. Ευχαριστούμε κύριε Τσίτσεστερ. κυρία Τζαβέλα. Επειδή πήρα θάρρος από αυτά που είπε ο Κλοντ Τούρμες, κύριε Επίτροπε, πράγματι είναι πολύ ακριβή η ενέργεια στην Ευρώπη και θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις ενδογενείς μας πηγές, είτε είναι shale gas, είτε είναι κάτι άλλο. Βλέπετε ότι και ο κύριος Τούρμες που εκπροσωπεί τους Πρασίνους εκφράζει τις ανησυχίες του για τις εισαγωγέ που κάνουμε σε πετρέλαιο και πρώτες ύλε από τρίτες χώρες. Ελπίζω ότι θα έχει και την υποστήριξή σας ε, των Πρασίνων πραγματικά για να αξιοποιήσουμε τις ενδογενείς μας πηγές και να μην έχουμε παράλογες αντιδράσεις από την πλευρά των, Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Επίτροπε και κυρία Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Τζαβέλα. Και τώρα η κυρία Τζόρνταν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο, διότι πραγματικά έχει ε, εξασφαλίσει αδιάκοπο διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα, Επίτροπε, που είπατε ότι χρειάζεται εξορθολογισμό τη πολιτική μα για την ενέργεια και ότι πρέπει να σκεφτούμε τον αριθμό των στόχων που θα θέσουμε εξακολουθώ να λέω ότι είναι υπερβολικά πολυάριθμοι στόχοι μας με ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καλύψουμε και άλλους δύο τομείς, την βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον και τις ανάγκες τους, δηλαδή ανταγωνιστικότητα και κοινωνικές πτυχές μαζί με το περιβάλλον και την αηφορία. Συμφωνώ με όσα είπε η κυρία Τζαβέλα, διότι θα πρέπει να συγκρίνουμε την τιμή της ενέργειας στην Ευρώπη με το τι συμβαίνει και το πώς διαμορφώνονται τιμές στις Ηνωμένε Πολιτείες. Έχουμε πολύ ψηλότερες ε, τιμές. Στην ε, πράσινη βλήβλο προβλέπονται συγκεκριμένε διατάξεις για την, ε, για την τιμολόγηση της ενέργειας. Και επίσης η άλλη ερώτησή μου είναι πώς υπολογίζετε να έχετε κατά νου κάποια εναλλακτική λύση θα έχουμε κάποια συμφωνία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών το 2015. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Τόμψεν για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ε, καλωσορίσω κι εγώ. Πραγματικά μας περάσατε πολλά μηνύματα, αλλά έχω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Είπατε ότι η ενέργεια θα πρέπει να είναι χαμηλών τιμών για να μπορεί ο καθένα να καλύψει τι ανάγκε του. Όμω έχουμε ενεργειακή ένδυα στην Ευρώπη πλέον. Οι τιμέ τη ενέργεια εξαρτώνται από το που ζει κανεί. Στο δικό μου διαμέρισμα στην Κοπενχάγη η θέρμανση είναι πολύ φτηνή ίσως και φτηνότερη από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Έχουμε λοιπόν τέτοια παραδείγματα στην Ευρώπη. Όμως πριν από τρεις εβδομάδες γίνονταν διαδηλώσεις ε, μπροστά στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο επειδή είναι πολύ υψηλέ οι τιμές της ενέργειας εκεί. Πέρυσι πήγα στην Ουγγαρία και με ρωτούσαν ε, οι ρωτούσαμε τους ανθρώπους ποιο είναι το σημαντικότερο πολιτικό ζήτημα και είπαν οι τιμέ τη ενέργεια στην Ουγγαρία 10% των φτωχότερων πολιτών δίνουν το 50% του εισοδήματό του για τη θέρμανση το χειμώνα. Πραγματικά λοιπόν θέλω να μου πείτε εάν μπορούμε να βρούμε αποτελεσματικέ λύσει εδώ. Τι θα κάνουμε για την ε, ενεργειακή ένδυα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή στρατηγική, είπατε κι εσείς, αλλά ειδικά για αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει ένας κοινό ορισμός. Τι θα πει ενεργειακή ένδυα καταρχάς. Εσείς δεσμεύεστε να ε, το προωθήσετε αυτό. Θα έχουμε μια τέτοια στρατηγική πριν το τέλος της θητείας μας. Διότι αυτό νομίζω ότι είναι το πλέον σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλω να σα ρωτήσω είναι τι γίνεται με την πράσινη βίβλο. Εξ κατάλαβα, είπατε σε ένα από τα σημεία της ομιλίας σας ότι η κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε δεσμευτικούς στόχους. Ιδάλω δεν θα δώσει αποτελέσματα. Είδαμε δεσμευτικού στόχου για το 2020, για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια δίνουν κάποια αποτελέσματα, αλλά η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν έδωσε αποτελέσματα. Τώρα θα έχουμε δεσμευτικούς στόχους μετρήσιμους για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα υπάρξουν ενεργεια... τέτοιοι δεσμευτικοί στόχοι στην πρότασή σας για το 2013. Μέσα μάλλον στη χρονιά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρόντι παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Πάντοτε χαιρόμαστε να συζητούμε μαζί σας. Εγώ πρόσφατα είδα ότι το σύστημα επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όγκο. Εδώ πήρατε μέτρα πρόσφατα για την δίληση των ορυκτών καυσίμων. Αυτό δεν αντιφάσκει με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερο ερώτημα. Γίνονται πολλές, πρέπει να γίνουν μάλλον πολλές επενδύσεις, προφανώς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά ακόμη δεν κάναμε λόγο για τους δημοσιονομικούς πόρους, τα κονδύλια. Κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο είναι υπέρ, συμπαρατάσσεται δηλαδή με αυτούς που υποστηρίζουν τα ευρωομόλογα τα Eurobonds. Έτσι μόνο θα εξασφαλίσουμε πόρους και κονδύλια τα οποία άμεσα να αποδοθούν για την ανακούφιση από την σημερινή οικονομική κρίση. Ιδιαιτέρως, εάν σκεφτούμε ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις για τις οποίες να μην μετανιώσουμε στο μέλλον. No regret. Και αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε κυρία Επίτροπε, έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε κύριε Πρόντι. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ, κύριε Επιτροπέ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη είναι, υπάρχουν πάρα πολλές ε, κρυφές επιδοτήσεις για την ε, παραγωγή ενέργειας από ορυκτές ε, πηγές, γι' αυτό είναι ευθύνη. Θα ήθελα να γνωρίζω τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σταματήσει αυτή η κρατική ενίσχυση. Και πώς σκοπεύετε να την τερματίσετε. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, το οποίο έχει μείνει πολύ πίσω στη χρηματοδότηση. Και υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, του να μελετήσουμε το εάν μπορούμε να έχουμε ένα έξυπνο δίκτυο και ένα υπερδίκτυο με άλλο τρόπο, ε, π.χ. μέσω των σιδηροδρομικών δικτύων. Τι γίνεται? Έχει σταματήσει αυτό, το ερευνάτε. Τέλος, συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε πως η επένδυση στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ο κατάλληλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια, όπως είπε η κυρία Τόμψεν, αλλά μήπως ο τρόπος είναι να είναι ο καθένας ο δικός του παραγωγός σε μικρή κλίμακα, ο παραγωγός ενέργειας. Έχετε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική που να τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Ε, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον Επίτροπο. Πάντοτε τον ακούω με ενδιαφέρον. Είναι ευφυής και έχει πρακτική προσέγγιση. Δεν είναι νέα που είναι στη δουλειά μας. Είπε δύο πράγματα που θέλουν τόλμη ότι δηλαδή, η ενεργειακή πολιτική δεν αφορά μόνο το διοξείδιο του ανθρώπου, όπω λένε και επίση, ότι δεν είναι ανταγωνιστικέ οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τώρα περνάμε από φάση ύφεση, χρειαζόμαστε απασχόληση, χρειαζόμαστε ανάπτυξη και χρειάζεται να είναι επομένω ανταγωνιστική και η ενέργειά μας. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος Τούρμες. Πολλά μπορεί να γίνουν όσον αφορά την δεσματικότητα στην ενέργεια. Μπορεί να γίνουν πολλά. Πολύ περισσότερο όπως θα κάνουμε τώρα. Παράδειγμα, στη δική μου χώρα, που λένε κελτικός τίγρης. Εκείνη την εποχή πληρώναμε ένα σωρό για το μαζούτ. Παρ' όλα αυτά, τα δημόσια κτίρια και τα νοικοκυριά θα πρέπει να πάμε σε κάποια μείωση για αυτά. Για όλους δηλαδή. 30-40% συνοφρατήρων κατανάλωση. Αυτό θα βοηθούσε. Άντε, ακόμα για να πάμε στο φυσικό αέριο παρόλα αυτά. Ε, έκανε για την Ρέτζη τη σχετική έκθεση και είπαμε ότι η υγειονομική ενέργεια ε, τέλος πάντων και με θαλάσσια έδατα μπορούμε να έχουμε παραγωγή ενέργειας για να είμαστε ανταγωνιστικοί που είναι πολύ σημαντικό. και πολλές εταιρείες του κλάδου να σας πούν ότι ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου πέρα από την Ευρώπη, στα διεθνή Για πέστε μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για το ότι σκέφτεστε και το μέλλον ε, και βεβαίως θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την Πράσινη Βίβλο και τις προοπτικές και την Ευρώπη του 2030. Έρχομαι στο πρώτο μου ερώτημα. Εάν σκεφτούμε πώς πρέπει να έχει το μέλλον, Mm. Σκεφτόμαστε και το παρελθόν. Είχαμε σε όλες τις χώρες ε, εθνικά μονοπόλια. Είχαμε ένα, δύο, τρία πακέτα απελευθέρωσης ε, της, της αγοράς ενέργειας και φαίνεται πως ε, με την αλλαγή των κανόνων πηγαίνουμε προς ένα σχεδιασμό της αγοράς, αλλά πάμε πάλι προς περισσότερη κρατική παρέμβαση. Οπότε κάπως προκλητικά να ρωτήσω. Παρόλη την απελευθέρωσή μας ε, απέτυχε η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτών. Ακολουθούσαμε μια πορεία που ε, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και μια άλλη παρατήρηση. Μιλήσατε για μεγαλύτερη σύγκληση ε, των διαφόρων μορφών ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης και είχαμε βέβαια σήμερα και την έκθεση Herbert Roll η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και διατύπωσε τις σκέψεις μας. Θα μπορούσατε να την σχολιάσετε. Οι ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζουν την πράσινη βίβλο της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Είπε ο Πίτροπος ότι μελετώνται οι τρεις βασικοί στόχοι. Τρεις ε, στόχοι ε, είναι αυτό που αναφέρατε ή αλλαγή της νοοτροπίας. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, διότι οι πολίτες μίλησαν για ενίσχυση των στόχων. Όμως, ίσως να έπρεπε να υπάρχει μια ιεράρχηση των στόχων. ένα πρωταρχικό και κάποιοι δευτερεύοντε. ε, για όλα αυτά που προτείνεται. Και έπειτα, μια και μιλάμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Μίλησε η συνάδελφο, για τι δημόσιε επιδοτήσει, για τον άνθρακα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν εδώ, τι άποψη έχετε, τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι δημόσιε επιδοτήσει, για τι κρατικέ επιδοτήσει, για τι πηγές, για τις Υπάρχουν εδώ προβλήματα σε κάποια μέλη με αυτού του είδου τι επιδοτήσει. Τι κάνει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε πει ότι μέχρι το 2020 θέλετε να καταργηθούν αυτές οι επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές. Εάν λοιπόν θέλουμε νέους στόχους, θα πρέπει να σκεφτούμε και την κερδοφορία. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα αυτές οι επιδοτήσεις να εξαλειφθούν πλήρως από, από την άποψη της κερδοφορίας. Έπειτα είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση για συνεργασία με ένα έγγραφο που μιλάει για εταιρική σχέση για την ενέργεια με τη Ρωσία. Σε αυτό το έγγραφο, σε αυτό τον οδικό χάρτη θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο με την ενέργεια και πώς αυτό συμβιβάζεται με την αδυναμία μας να προθίσουμε παρκώ το τρίτο πακέτο για την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστούμε, κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σήμερα έχουμε μια δεύτερη μελέτη για τα τεχνολογικά προβλήματα των ε, βελγικών πυρηνικών εργοστασίων στο Ντόλ και στο Τιάνος. Και το πρόβλημα είναι πως ακριβώς τέτοια προβλήματα δεν καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά τεστ κοπόσεως, αλλά υπάρχουν. Και τώρα φαίνεται πως ε, κατά τη διάρκεια της ε, κατασκευής του τυράνζ υπήρχε ένα πρόβλημα με κάποιον χαλίβδινο δακτύλιο που θα πρέπει να αλλάχθεί. Και Βεβαίω ε, σήμερα αξιολογούμε διαφορετικά την ασφάλεια από την εποχή που χτίστηκε ε, το εργοστάσιο αυτό. Οπότε σκοπεύετε στο προσεχές μέλλον να αναθεωρήσετε την οδηγία για τις ε, προδιαγραφές ασφαλείας των πυρηνικών εργοστασίων. Και το δεύτερο ερώτημα, αναφερθήκατε στην ασφάλιση των πυρηνικών εργοστασίων για την αστική ευθύνη που θέλετε να θίξετε ξανά. Είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα γιατί θεωρώ πως οι κίνδυνοι ε, που υπάρχουν και βλέπουμε στο Βέλγιο αξιολογούνται και θα ε, είχαν αξιολογηθεί τελείως διαφορετικά εάν ο διαχειριστής ε, ήταν ε, υπεύθυνο, είχε την πλήρη αστική ευθύνη σύμφωνα με την αρχή Ριπένον πληρώνει. Πότε λοιπόν μπορούμε να αναμένουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επιτροπέ στην Επιτροπή Ήτρε. Στα τέλη Νοεμβρίου η Επιτροπή αυτή υπερψήφισε τη δέσμη μέτρων για το Horizon 2020. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα ψηφίσαμε ομόφωνα. Με φιλόδοξους στόχους για να αντιμετωπιστούν ενεργειακές προκλήσεις. Αυτό σημαίνει ένα υψηλότερο ποσοστό από τον προπολογισμό. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν ο τελικό αριθμό για το Horizon 2020, Όμω αυξήσαμε το μερίδιο τη ενέργεια στους συνολικού στόχου του Horizon 2020. Και νομίζω ότι είναι ευρύτερο το θέμα, θα έπρεπε περισσότερα να καλύπτονται και να είμαστε κι εμεί πιο φιλόδοξοι και στην ενεργειακή υποδοτικότητα από ό,τι στην αρχική πρόταση και στο κεφάλαιο για την αποθήκευση για τα FE δίκτυα, το CCF και το CCU. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση της του ενεργειακού προστατευτισμού και της προστασίας καθώς και να δούμε τι θα γίνει με την ευφυή ενέργεια για την Ευρώπη και το σχετικό πρόγραμμα. Θέλουμε να γίνει έρευνα και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, τα νέα αυτά σημεία δεν έχουν γίνει ακόμη αποδεκτά. Υπολογίζουμε σε εσά λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εντατικές σας ε, προσπάθειες και διαβουλεύσεις. Επηρεάστε την τελική απόφαση, να γίνει κάτι καλό για την ενέργεια. Νομίζουμε ότι ω τώρα όσο έχουμε συμφωνήσει είναι ισόρροπα και πολύ εύστοχα. Επίση, ένα τελευταίο σχόλιο είπατε ότι ανησυχείτε για το τελικό αποτέλεσμα για την ε, εφταετία, για το Horizon 2020 όμως ε, φαίνεται να έχουμε βασίσει και όλες μας τις ελπίδες. Τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα από το Συμβούλιο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και σχέσεις συνεργασίας με τα διαρθωτικά ταμεία. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να αντιδράσουν τα κρατημέλη. μελη Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση ο κ. Σοντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την άριστη παρουσίαση που μας κάνατε για την ενεργειακή μας πολιτική. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, οι επιπτώσεις των ατυχημάτων. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι στην αλυσίδα της αντίδρασή μας να λαμβάνονται υπόψη και για τα υδροελεκτρικά και για τα γεωθερμικά και για την πυρηνική ενέργεια το τι μπορεί να γίνει με τα ατυχήματα. Ξέρετε επίσης τι γίνεται με τα κονδύλια και πώς μπορεί να κινητοποιηθούν αυτά. Το είδαμε πρόσφατα με το πετρέλαιο. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες περιστάσεις, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει. Επίσης, για τα ύδατα. Έχουμε ε, δημιουργήσει ένα μοντέλο όπου υπάρχουν λίγα κέντρα παραγωγής και πάρα πολλά σημεία κατανάλωσης. Πρέπει να πάμε τώρα προς ένα μοντέλο που θα υπάρχουν πολλά σημεία παραγωγής να πολλαπλασιάζονται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ιδίως. Πώς βλέπετε λοιπόν το θέμα των δικτύων θα μπορούσε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εταιρεία για τα ενεργειακά δίκτυα. Προφανώς αυτό δεν συνάδει με την ε, νοοτροπία και την κουλτούρα του ΕΛΚ, όμως εσείς πώς βλέπετε το θέμα των δικτύων και τη χρηματοδότησή τους και για την νομοθεσία. Τρίτη παρατήρηση. Είπατε θα κάνουμε νομοθετική πρόταση στο τέλος της χρονιάς. Ειλικρινώς μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε γιατί έχουμε και εμείς την υποχρέωση να ετοιμαστούμε για τις ευρωεκλογές θα αποφασιστούν πολλά με τι ευρωεκλογέ του 2014. Εντάξει για την πράσινη βίβλο, εντάξει για τι προτάσει ανακοινώσεων που κάνατε και ε, τι πρωτοβουλίε που προτείνατε. Όμω, α περάσουν και ευρωεκλογέ ώστε να ε, εγκρίνουν από νομοθετική άποψη το νέο Κοινοβούλιο και, ε, το νέο συμβου... και η νέα Επιτροπή του στόχου του 2020 που δικαίω ε, του τονίσατε και του θυμήσατε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε τον κύριο Ντί. Κύριε Επίτροπε, έχετε να απαντήσετε σε ένα σωρό ερωτήσει. 15 λεπτά. Herr Turmes hat einen Schwerpunkt auf der Analyse der Energiepreise gelegt. Ο κύριος αναφέρθηκε στις τιμές της ενέργειας. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Γεγονός είναι πως η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις τιμές του πετρελαίου. Και η τιμή του πετρελαίου δεν θα πέσει από ό,τι φαίνεται. γεγονό είναι πω αυτή τη στιγμή είναι ευθυνότερο ο άνθρακα για ένα απλούστατο λόγο. Οι Αμερικανοί ε, μέχρι στιγμή ε, έκαιγαν άνθρακα, τώρα έχουν ε, αέριο, έχουν λοιπόν περισεβούμενο άνθρακα, τον εξάγουν στην Ευρώπη και είναι ευθυνό για, τις, για την παραγωγή ενέργειας, για θέρμανση και ηλεκτρισμό. Η τιμή του πετρελαίου όμως ανέβηκε ε, γιατί είναι μια, ε, ε, μιλάμε για την παγκόσμια αγορά. Μεταξύ αμερικανικής και ευρωπαϊκής αγοράς υπάρχει μια διαφορά γύρω στο 10% που δεν υπήρχε. Που προέκυψε μέσω της παραγωγής της εσωτερικής των ΙΠΑ από άμμο και διάφορες άλλες πηγές από την την εγχώρια παραγωγή. Αλλά το, το 10% αυτό στον παγκόσμιο ανταγωνισμό δεν ξέρουμε αν είναι. δεν είναι ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα. Δηλαδή στο Σικάγο, στη Σανγκάη και στο Ρότερνταμ ε, οι τιμέ είναι ίδιες ε, όταν μιλάμε δηλαδή για την θέρμανση, για τους βιομηχανικούς πελάτες, για τη χημική βιομηχανία, για οτιδήποτε. Αλλά ακριβώς αυτό δηλαδή μία τιμή στην παγκόσμια αγορά του πετρελαίου, ανεξάρτητος του ύψους της, η οποία δεν θα επηρεάζει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, δεν υπάρχει για φυσικό αέριο και ρεύμα. Υπάρχει για τον άνθρακα και όταν θα τελειώσει το 2018 η ενίσχυση του άνθρακα και ε, αυτή τη στιγμή δεν το έχει κάνει κανένας ε, κράτος μέλος, θα συνεχίσει να υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή η ενίσχυση από καθαρά εθνικά κονδυλιά. Η Γερμανία, παραδείγματο χάρη η χώρα μου, αυτή τη στιγμή αποδέχεται κάτι τέτοιο. Το αποδέχονται όλα τα κόμματα. Το θέμα λοιπόν φαίνεται πως ε, είναι ανοιχτό σε κάποιες κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες και στην ε, Ισπανία. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει μία παγκόσμια αγορά και τιμή. Ε, ανεξάρτητος το αν μιλάμε για, τον Καναδά, την Αφρική ή οπουδήποτε. Και βεβαίως πάνω σε αυτό προστίθεται και η τιμή των μεταφορικών. Οπότε αν θέλετε, έχουμε κάποιους ίσους ανταγωνισμού. Το ίδιο για την βιομάζα, ε, υπάρχει μια κάποια ιονή παγκόσμια αγορά, για το ουράνιο το ίδιο, αλλά όχι για το φυσικό αέριο, όπως σας είπα, και τον ε, ηλεκτρισμό. Έχουμε αφενός για λόγους ε, το σχιστολιθικό αέριο το οποίο αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε ένα 25% της μέσης τιμής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως δεν ξέρω αν θα παίξει το σχιστολιστικό αέριο τον ρόλο που έχει παίξει στη ΣΥΠΑ για πολλούς λόγους. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω την επιλογή αυτή να μην την απορρίψετε γενικώ. Θα μπορούσαν κάποιες χώρες να το κάνουν. Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία. Ίσως οι Βαλτικές ίσως κεντροευρωπαϊκές χώρες γενικώ. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν με αυτή την επιλογή. Άλλες αυτή τη στιγμή είναι κατά γενικώ, η Γαλλία. Αλλά, σας λέω, από τις συνομιλίες με τους Ρώσους εταίρους μας, ακόμα και η επιλογή αυτή τους προξενεί νευρικότητα. Γιατί η δική τους λογική είναι αέριο από τη Ρωσία, αγωγή από τη Ρωσία, μακροπρόθεσμα συμβόλαια, έτσι. Και πληρώστε ούτω ή άλλω. το θέλετε ή δεν το θέλετε, και σύνδεση με την τιμή του πετρελαίου. Ε, δεν θα στέκουν όλα αυτά εάν περάσει το ε, σχιστολιθικό αέριο στις αγορές spot και εάν έχουμε και ε, τέρμινα λιγροποιημένο φυσικό αέριο. Οπότε θα μπορέσει να μας βοηθήσει τουλάχιστον για καλύτερες συνθήκες διαπραγμάτευση με τους Ρώσους και για δική μας παραγωγή αέριου. Και... Παρόλα αυτά είναι σαφές πως δεν θα επιτύχουμε τις τιμές των Αμερικανών. Αλλά το ζήτημα μεσοπρόθεσμα είναι ε, θα κοστίζει το αέριο στην Ευρώπη το τετραπλάσιο όπως κάνει τώρα ή το μισό ή το εξαπλάσιο. Ε, δεν πρέπει τουλάχιστον να αυξηθεί αυτή η διαφορά της τιμής. Εντάξει, να δεχτούμε κάποια διαφορά, αλλά όχι όποια να είναι. Έτσι. Γιατί έχουμε και το, ε, το εργατικό κόστος. Είναι ένα ανάλογο ερώτημα. Δεν θα γίνουν χώρες φτηνής εργασίας οι ευρωπαϊκές χώρες. Ε, αλλά όταν τη συγκρίνουμε με την Μαλαισία, μιλάμε για τιμές ε, δεκαπλάσεις. Οπότε εδώ πέρα θα παίξει ρόλο η ε, ακρίβεια ή η ποιότητα κτλ. Οπότε μπορούμε να αποδεχτούμε το υψηλότερο κόστος και στην εργασία και στην ενέργεια, αλλά όχι όσο μεγάλη είναι και να είναι αυτή η διαφορά. Και για το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή προτείναμε στο Συμβούλιο μια σύγκριση των τιμών της ενέργειας. Έχουμε τεράστιε διαφορές στην Ευρώπη τη ηλεκτρική και αυξάνεται η διαφορά με χώρες ε, αραβικές, με τη ΣΥΠΑ και σε άλλες περιοχές. Και είναι σαφές πως το ρεύμα είναι όλο και πιο σημαντικό για τη βιομηχανία. Βεβαίω, πράγματι, η κατά μέσο όρο το κόστος του ρεύματος είναι 3 με 4% του τζίρου της βιομηχανίας. Αλλά καταλαβαίνετε πως έχουν το... Τι λέμε μέσος όρο, δηλαδή όταν ε, το ένα πόδι είναι στο φούρνο και το άλλο στο ψυγείο λέμε μέσος όρο θερμοκρασίας είναι 20 βαθμοί, δεν είναι έτσι. Έτσι αυτή τη στιγμή είναι σημαντικότερο το κόστος του ρεύματος από ότι το κόστος εργασίας. Ειδικά όταν μιλάμε για βιομηχανίες όπως ε, αλουμίνιο, άνθρακας, ε, χαρτί, χαλκός, ενεργοβόρες δηλαδή. Και μην ξεχνάτε, θα... Κύριε Τούρμε, κύριε Τούρμες, έχουμε και αυτή την αλυσίδα τροφίμων την έτικα στην, ε, στην Γερμανία. Όχι, μην το, είναι θέσει εργασία οι οποίε χάνονται. Έτσι. Γιατί εσείς λέτε όχι, θέμε μόνο τις νέες θέσεις εργασίας. Και δεν χρειαζόμαστε τις καινούριε. Τι παλιέ, με συγχωρείτε. Όχι, τι χρειαζόμαστε όλε. Και τι παραδοσιακέ και τι καινούριε. Μα, κυρία Χάρμ, ε, μπήκατε λίγο αργά. Είχα απαντήσει στην ερώτησή σα. Μπήκατε λίγο αργά στην αίθουσα. Είχα απαντήσει την, ε, την ερώτηση, ήρθατε και την επαναλάβατε. Εντάξει. Ε, αν είχατε. Μα Α σεβαστούμε και, την άποψη του άλλου, έτσι. Πρέπει να τις διατηρήσουμε όλες, όλες τις θέσεις Έχει λοιπόν η ευρωπαϊκή χαλιβουργία και προβλήματα προξένησε μόνη τη, αλλά και το πρόβλημα της τιμής ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι ο στόχος μας και μετά να ακολουθήσουμε μια ανάλογη ενεργειακή στρατηγική, όχι με την ενεργειακή στρατηγική να διώχνουμε τις βιομηχανίες. Και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Αναμένω την απόφασή σας με σεβασμό. Εγώ είμαι υπέρ του backloading, αλλά μια τέτοια παρέμβαση με 900 εκατομμύρια μονάδες απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή Βιομηχανίας, στην ΔΕ Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, έγινε δεκτή και λέγαμε ε, το πολύ μία φορά θα γίνει. Άπαξ. Βλέπουμε λοιπόν για τεράστια αλλαγή του πολιτικού κλίματος. Γιατί πριν από πέντε χρόνια θα λέγανε backloading, όχι, είναι πάρα πολύ λίγο, πρέπει να κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερα. Και στο Συμβούλιο δεν είναι ε, μόνο βουλευτές. Εκπροσωπούνται, μην ξεχνάτε, πως είναι μέλη των ε, κυβερνήσεων, των συνδικάτων, τον πάνω και λένε έχουμε το 2003 στόχους κλιματικούς και στόχους ενεργειακούς και στόχους αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας. Και όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και σε πάρα πολλές χώρες άλλες μας λένε, κοίτα, παράτα μας ήσυχους τώρα με όλα αυτά. Ισπανία, Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ελλάδα έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν θέλουν να τα ξανακούσουν αυτά τα πράγματα. Και πίσω από τους Πολωνούς κρύβονται Σλοβάκοι, Τσέχοι, Βαλτικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία. Και χαίρονται που οι Πολωνοί με τους μεγάλους τους ώμους προβάλλουν το βέτο και έχουν τις πλάτες να το κάνουν. Έτσι, εγώ είμαι υπέρ της συνέχισης αυτής της υπόθεσης μέρα από το 2020, αλλά πρέπει όλοι, εμείς, εσείς και το Συμβούλιο, να είμαστε ρεαλιστές και να μην κατακαιρματίσουμε τελείως και καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή πολιτική του κλίματος. Δεν θα χρειαζόμαστε μετά επίτροπο κλίματος και ενέργειας και ούτε διαβουλεύσεις εδώ μέσα. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλοι λίγο να χαλαρώσετε λίγο τις απαιτήσει σας. Και το backloading είναι ένα ε, μήνυμα εδώ πέρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο έχει προξενήσει φοβερό αντίκτυπο στο Συμβούλιο. Τώρα, ε, με ρωτήσετε γιατί εθνικές παρεμβάσεις. Οι ανανεώσιμες πηγές χρειάζονται κρατική επιδότηση, άμεση ή έμεση. Βλέπουμε πως ε, η αιωλική στην ξηρά πλησιάζει στην αγορά η αιωλική στην θάλασσα εξακολουθεί να χρειάζεται κρατική ενίσχυση. Η γεωθερμία, η ενέργεια στη θάλασσα χρειάζεται ακόμη πολύ περισσότερο χρόνο και δεν θα μπορέσει να υπάρξει χωρίς κρατικές ενισχύσεις. Τα φωτοβολταϊκά ακόμη χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο με κρατικές επιδοτήσεις. Έχουμε επίσης Ε, ξαφνικές απότομες αλλαγές επί το χείρο της Ευρωπαϊκή, των ευρωπαϊκών νομοθεσιών για την επιδότηση. Πρέπει οπωσδήποτε οι επιδοτήσεις σταδιακά να μειωθούν και κάθε πηγή ενέργειας να μπει στην αγορά. Και αυτό το οποίο έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες νομίζω ε, προκαθορίζουν το τι θα γίνει στο μέλλον. Τώρα, με ρωτήσετε τι θα γίνει μέχρι το φθινόπωρο και τι... γιατί πρέπει να είναι προετοιμασμένο το Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα έχουμε την οδηγία πυρηνική ασφάλεια, την πρότασή μα δηλαδή, τον Μάιο, κάτι το οποίο μα ζητήσατε. Το φθινόπωρο θα έχουμε την πρότασή μα για την κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και την υποχρέωση ασφάλειας και έχει δίκιο ο κύριος Τούρμες, το θέμα είναι τι, τι ορίζουμε ως ζημία ποιο είναι το φάσμα της υλική ζημιάς, της ζημιάς στον άνθρωπο, στην ε, ιδιοκτησία και στη φύση. Εγώ θέλω να το επεκτείνω στο μέτρο του δυνατού. Αλλά θα σας πω το εξής. Είχα ήδη κάτι άτυπες συζητήσεις στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν το βλέπω διατεθειμένο να δεχτεί μεγάλα άλματα. Για πολλούς λόγους. Και ο βασικός λόγος βεβαίως είναι πως είχαμε το ψήφισμα 13 κρατών μελών που το κατέδειξε. Είχαμε τα 13 πυρηνικά κράτη-μέλη πλην της Γερμανίας που συναντήθηκαν και ο βασικός λόγος είναι, ε, μας είπαν δηλαδή, δεν θέμε να ανακατευτούν οι Βρυξέλλες σε αυτό. Και εδώ πέρα προσπαθώ να βρω έναν συμβιβασμό. Αλλά όσο πιο μαξιμαλιστικές θέσεις έχουμε, τόσο πιο πολύ θα μας πούνε στο Συμβούλιο, κοίτα, δεν έχετε ε, καμιά δουλειά σε όλα αυτά. Δηλαδή εμεί θα έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αλλά αυτά θα πάνε κατευθείαν στο αρχείο, έτσι. Δηλαδή το να αναγνωρίζουμε και ποια είναι τα όρια μας είναι νομίζω εξίσου σημαντικό και να προτείνουμε εφικτά πράγματα από το να προτείνουμε μεγάλα βήματα και να μην αλλάξει τίποτα τελικά έτσι. Έχουμε λοιπόν επίσης την πρόταση PCI, δηλαδή ποια είναι αυτά τα, τα έργα τα οποία θεωρούμε κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, διασυνδέσεις, ε, δίκτυα, ε, τέρμινα λιγροποιημένο φυσικό αερίο κτλ. Ενεργειακή έμβια. Και εδώ πέρα θα ε, υποβάλουμε την πρότασή μας. Το αποφασιστικό είναι το εξής. Ενεργειακή έμβια. κινητικότητα, αλλά και θέρμανση, ψήξη και ρεύμα είναι αναμφισβήτητα. Και ομολογώ, συζητάμε συχνά για ε, το ηλεκτρικό ρεύμα και όχι αρκετά για τη θέρμανση, παραδείγματος χάρη. Το αποφασιστικό ερώτημα είναι, θέλουμε να την μειώσουμε μέσω ε, δωρεάν, μείωση με την ενεργειακή φτώχεια μέσω δωρεάν παροχής ενέργειας ή χαμηλών τιμών ή να, μπουν σε ένα να μπει σε ένα καλάθι κοινωνικών παροχών και η ενέργεια. Εγώ είμαι υπέρ του δεύτερου για να μην έχουμε παρέμβαση στην αγορά. Δηλαδή μετά τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο δωρεάν ψωμί, στη ε, δωρεάν αναψυχή, στη δωρεάν εφημερίδα τι θα, θα έχουμε έναν προϋπολογισμό, ένα επίδομα εάν θέλετε, το οποίο θα πηγαίνει και θα καλύπτει από αυτό ο κοινωνικά ασθενέστερος ε, πιθανώς ε, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, ε, μια κινητικότητα κτλ. Και όχι να παρέχει τα αγαθά το ίδιο το κράτος. Αλλά για το πετρέλαιο και τα προϊόντα τα οποία όπως σας είπα είναι προϊόντα των διηληστηρίων. Πρέπει να διηλίζονται στην Ευρώπη και να μην τα παίρνουμε έτοιμα διηλισμένα από τη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί πρόκειται και για θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στα διηλιστήρια. Επίσης κύριε Πρόντι αναφερθήκατε στα ευρωομόλογα. Εγώ θα τα έλεγα ε, ομόλογα έργων. Τέλος αν δεν δικιά μου δουλειά. Αυτή είναι του κυρίου Ρεν αλλά για τα ομόλογα έργων τα ζητάμε. Ε, αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες απόπειρες και αν έχουμε το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη βλέπετε πως δεν έχουμε επιδοτήσεις ε, άμεσες μετρητών γιατί έχουμε 35% Έχουμε εγγυήσεις και ομόλογα έργων στην περίπτωση αυτή. Και έτσι μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε το ποσό που θα διατεθεί για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών ε, υποδομών. Μετά είχαμε το ερώτημα τι γίνεται με τους Ρώσους εταίρους μας. Πέμπτη Παρασκευή πάλι έχουμε τη συνάντησή μας στην Μόσχα. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Οι Ρώσοι δεν δέχονται τα πακέτα μας για την εσωτερική αγορά. Δηλαδή, το, την πρόσβαση τρίτων μερών και την ε, αποδέσμευση. Θέλουν μια συμφωνία πως η αγωγή του φυσικού αερίου ειδικά που έχουν φτιάξει οι Ρώσοι να έχουν μια γενική εξαίρεση από την πρόσβαση τρίτων μερών και την ιδιοκτησιακή αποδέσμευση. Δεν είναι δυνατό. Οι κανόνες μας είναι ισχύον δίκαιο, πρέπει όλοι να τους δεχτούν. Ε, Νορβηγία, Αλγερία, οι εταιρείε της Ένωσης και, και η Gazprom. Και βεβαίως γνωρίζουμε πως έχουν και ανταγωνιστές και η Novatec και η Rosneft που παράγει και εξάγει κυρίως πετρέλαιο θέλει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του αερίου και να στείλει ε, LNG στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί την ε, Gazprom. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε έτσι ανταγωνισμό. Και πιθανώ να μπορέσουμε και να εξάγουμε και στη Ρωσία, όχι μόνο να έχουμε προ μία κατεύθυνση τη ροή. Τώρα, για τον ορίζοντα 2020, το εάν θα είναι 60, 70 ή 80 δισεκατομμύρια τα κονδύλια πρέπει να ορίσουμε οπωσδήποτε και τις προτεραιότητες μας, αλλά να είστε σίγουροι πως στην πρόταση προϋπολογισμού για την ε, ενέργεια και την ε, έρευνα στον τομέα της ενέργειας θα έχουμε οπωσδήποτε αρκετά μεγάλη χρηματοδότηση. Και διάβασα με ευχαρίστηση τις προτάσεις του ε, Κοινοβουλίου και νομίζω πως ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία ήθελε η Κομισιόν σχεδόν 100%. Τώρα, για Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας μιλήσατε. Ακούγεται ωραίο. Αλλά κάποιοι λένε πως τα δίκτυά μας και η αγωγή πρέπει να αναπτυχθούν κάπως ε, έτσι, κεντρικά. Εντάξει, το ποιο είναι το υπόδειγμα, η Κίνα. Που υπάρχει μια εταιρεία και κανονίζει τα πάντα. Αλλά είμαι ρεαλιστής Βεβαίω, Τα κράτη-μέλη δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο. Δεν θα δώσουν τη δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό υπάρχουν δύο δυνατότητες. να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος συντονισμός και εναρμόνιση. Αυτά είναι λοιπόν τα μέσα που έχουμε στην περίπτωση, στην διάθεσή μας για να επιτύχουμε όσο περισσότερα μπορούμε, γνωρίζοντας τις εθνικές και περιφερειακές διαφορές και τα συμφέροντα που είναι κατά ε, πανευρωπαϊκών δικτύων και υποθέτω πως θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Αναφέρατε επίσης ε, τα πυρηνικά εργοστάσια και πράγματι έχετε δίκιο, εμείς εξετάσαμε βλάβες που προέρχονται από κάποια εξωτερική ε, παρέμβαση. Τώρα κακοτεχνίες στην κατασκευή ε, δεν τα είχαμε υπολογίσει. Το τι είχαν κάνει δηλαδή οι Βέλγοι πριν από τόσα χρόνια και ε, σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν όσον αφορά τις επισκευές, δεν το ξέρουμε, αλλά οπωσδήποτε ε, βασιζόμαστε στην ε, ποιότητα και την αντικειμενικότητα της βελγικής ρυθμιστικής ε, αρχής και του βελγικού ε, κράτους. Γιατί υπάρχει, όπως είπα, αυτή η επικουρική δομή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο και για την παρουσία του εδώ σήμερα και επειδή απήντησε δείξω δικά σε όλε τι ερωτήσει που του τέθηκαν. Ευχαριστούμε Επίτροπε και το επανειδήν. Να συνεχίσουμε τώρα. Έχουμε ένα τέταρτο καθυστέρηση. Αλλά επειδή είμαστε ευφιέστατοι θα ε, αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο. Ο κύριος Βιντάλ κουάντρα, τώρα εισηγητή για την ποιότητα των καυσίμων και τι οδηγίε σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ. Ο κύριος Βιντάλ Κουάντρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα. Να πω τα καλύτερα για την κυρία Λεπάζ που είναι η συγκεκριτή της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ήταν σε επαφές μας ε, ε, ό,τι καλύτερο τόσο να μπορούσαμε να συντονιστούμε οι δύο επιτροπές. Καλώς όρισες κορίνού εδώ στην Εδρίαση. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα ξεκινούν οι συζητήσεις στην Επιτροπή μας. Αφορούν αυτή την πρόταση. Σε σχέση με το τι θα κάνουμε, με κάποια επίμεχα ζητήματα και εύχομαι να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό προνομαστή. Στόχος της προτάσεως, είμαι βέβαιος ότι συμφωνούμε με αυτού, ο στόχος είναι πάρα πολύ θετικός είναι το τι θα κάνουμε με την αλλαγή της χρήσης της γης σε σχέση με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις υπάρχουσες αγροτικές γέες. Πώς θα χρησιμοποιηθούν για να παραγάγουμε ε, βιοκαύσιμα. Τώρα, υπάρχει τέτοια μετακίνηση σε νέες γέες που δεν χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή προηγουμένως για σκοπούς γεωργικούς όπως ας πούμε ε, λιμόνες και δάση και οπότε τώρα χρησιμοποιούνται αυτά τα εδάφη για βιομάζα. Έτσι όμως έχουμε απόλυτη έχουμε ζημιά όσον αφορά τη βιοπικιλότητα και έχουμε και αύξηση των βαρερών εκπομπών. Να δούμε τώρα επόμενος πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη μείωση των ε, του, του, του, άνθρακο, γιατί είναι πάγια πολιτική πολιτική Ένωση, δεν μπορεί να γνωρίσουμε παρόλα αυτά. Αυτά τα μέτρα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα ε, προτείνει προκαλούν κάποια ερωτηματικά. Έχουμε τρία βασικά ζητήματα τα οποία αξίζουν τι προσοχέ μα. Πρώτα-πρώτα, κάποιου παράγοντε. Παράγοντε όπου προσάπτουν συνδέουν με αυτό το σύστημα iLook κάποιον συντελεστή σε κάθε προϊόν, σε κάθε φυτό για τις εκπομπές. Αυτό το λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά όμω οι απόψει των ε, επιστημόνων σε σχέση με αυτούς τους ε, ε παράγοντε δεν ε, ε καταλήγουν σε κάποια ομοφωνία. Επομένως το iLook είναι δυνατόν, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και σταθερά. Και επομένω αυτή η αξιολόγηση από τη βάση των παραγόντων, των συντελεστών του ILOC ε, επιβάλλει τον υπάρχει κάποιο είδου ε, οικονομικό μοντέλο το οποίο να διέπει τη χρήση του, γιατί πάντα με τα πρότυπα αυτό γίνεται. Αυτό το μοντέλο μα ε, μας οδηγεί σε κάποιο είδου περιορισμού σε κάποιο είδου αβεβαιότητε. και επομένω είναι πάρα πολύ λογικό να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο νομοθέτημα δεσμευτικό ε, για να ρυθμίζει αυτούς τους συντελεστές ε, επί των οποίων υπάρχει τόση διχογνωμία. Θα πρέπει επομένω περιοδικά να γίνεται μια ενημέρωση, μια επικαιροποίηση αυτών των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται, των κριτηρίων. Και αυτό θα αφορά την νομοθεσία. Τι θα πρέπει να είναι νομοθεσία, θα πρέπει να είναι προβλέψιμη και να είναι και σταθερή. Τώρα το δεύτερο σημείο αφορά το κενό, αυτή τη διαφορά του 5% όσον αφορά την ε, μετατροπή ε, το, το, το, της ε, συμβατικής παραγωγής. Αυτό θέλουμε να περιοριστεί και να μπορέσει να μείνει στα ε, σημερινά επίπεδα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες επενδύσεις, αυτές οι οποίες έχουν συντελεστεί, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το 10%, το 10% του στόχου που έχουμε στις μεταφορές για το 2020 όσον αφορά τα ανανεώσιμα. Και αυτό είναι μια πρόβλεψη, είναι ένας κανόνας Δεσμευτικό. Το θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη μάλλον δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτό το στόχο εάν ε, έχουμε αυτή τη διαφορά η οποία θέλουν να επιβάλλουν. Γιατί ε, έχουμε τα ηλεκτρικά οχήματα ω εναλλακτική στα ανανεώσιμα και τα οποία μα δίνουν περισσότερη αποτελεσματικότητα στο του κινητήρε. Δεν θα είναι αρκετά όμω τα ηλεκτρικά οχήματα τόσο ώστε να μπορέσουμε να άρουμε αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί να το πληρώσουν τέλο πάντων. Γιατί θα πρέπει να δούμε ότι δεν θα έχουμε κάποια δυσμενή διάκριση, γιατί έχουμε ακριβώ διαφοροποιημένη διαφοροποιημένα αποτελέσματα σε αυτά τα κριτήρια Αιλού. Άρα ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πάντως και τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη τη υπαίθρου. Τώρα, η Επιτροπή λέει στα κρατημένα θα πρέπει δύο φορές ή και τέσσερις φορές να υπολογίσουν τα βιολογικά καύσιμα σε σχέση με το εάν τηρούν, εάν συμμορφώνονται στον στόχο του 10%. Αυτό τι είναι. Είναι κίνητρο όσον αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ή καταλήγει να είναι ε, ένα κόλπο μαθηματικό το ώστε τα κρατημέλη τεχνητά να παρουσιάσουν, να εμφανίσουν τήρηση του στόχου είναι επομένως δίκοπο μαχαίρι. Γιατί έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε αντικίνητρο για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Άρα χρειάζεται ένα προβληματισμός ει βάθο. Για το κατά πόσον είναι δόκιμα τέτοιο μέτρο. Το βασικό μέσο πολιτική είναι αυτοί οι δείκτες. Μας οδηγούν στο να διαπιστώσουμε τι έχουμε καταφέρει για να μειώσουμε τα, τις εκπομπές τις βλαπτικές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να υπάρξει ανάπτυξη σε βιομηχανία και γεωργία. Άρα, η σωστή προσέγγιση είναι η σφαιρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα για να ε, λάβουμε υπόψη το ILUC αλλά θα πρέπει να διαλέξουμε εκείνα τα μέτρα τα οποία θα οδηγούν στα όσο γίνεται λιγότερα αντικίνητρα παραγωγής βιοκαυσίων. Τα μέτρα εκείνα τα οποία δεν θα εμφανίζουν δυσμενείς συνέπειες για τη βιομηχανία, ιδίω με τους σημερινούς καιρούς τη κρίση. Άρα χρειάζεται κάποιος επιμέρους στόχος για τα προχωρημένα βιοκαύσιμα. Πώς θα μπορούμε έτσι να έχουμε λίγο τις εκπομπές αυτά τα προχωρημένα βιοκαύσιμα που δεν τα έχουμε σήμερα. Έτσι θα τονώσουμε, θα δώσουμε κίνητρο για την παραγωγή. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι μέρους στόχοι θα έχουν ως ορόσημο μια χρονιά, μια καταληκτική ημερομηνία μετά το 2020. Επίσης να έχουμε κάποια μέτρα μετριασμού όπως παραγωγή σε υποθυσμένες γέες ή υπαχρησιμοποιητές. Εκεί να παραγαγούμε δύο καύσιμα. Εν κατακλείδη. Δηλαδή τελειώνω, τελειώνω θέλω να σας πω, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένα δίλημα. Το εξή. Δεν είναι εύκολο να γίνει τώρα η επιλογή. Είτε θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό το 10% στόχο σε ενέργεια, σε μεταφορές και εκεί έχουμε αυτή την πρώτη της Επιτροπή για πολλαπλό υπολογισμό ή θα πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε τον κανόνα του ΑΕΛΟΚ χωρίς να περιορίσουμε όμως την παραγωγή μας για τα δύο καύσιμα πρώτης γενιάς. Εγώ έτσι βλέπω τα πράγματα. Όπως βλέπετε, δεν είναι αυτονόητα τα πράγματα. Άρα, θα πρέπει με πνεύμα εργασίας να συνεργαστούμε και να ξέρουμε μια λύση. Περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις απόψεις σας. Όλων τις απόψεις γιατί τις απόψεις των ε, σχεδόν εισηγητών. Τις ξέρω μια που είχαμε μια τέτοια θετική παραγωγική ανταλλαγή απόψε. Θέλω να μου πείτε τι πρεσβεύετε για όλα αυτά και να μου πείτε και τι άλλο πρεσβεύετε για ό,τι άλλο σκεφτείτε σχετικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βινταλ Κουάντρα. Για τρία λεπτά η κυρία Τόμψεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. για τον τομέα των μεταφορών και τον τομέα της ενέργειας ξέρουμε τη σημασία των ορεικτών καυσίμων και τη βαρύτητά τους. Είναι τεράστια σημασία σε αυτό. Μιλήσαμε μόλις τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση των τιμών. Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιλέξει έναν βιωσιμότερο τομέα και για τις μεταφορές και για την ενέργεια. Πιστεύω ότι τα βιοκαύσιμα και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν είναι ένας τρόπος να απαλλάξουμε από τον τομέα των μεταφορών τομέα μεταφορών από τα όρυκτα καύσιμα. Θυμάστε ότι ο στόχο των 10% που αποφασίσαμε δεν είναι 10% βιοκαύσιμα, αλλά 10% ανανεώσιμα καύσιμα στον τομέα των μεταφορών. Εξού και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλε δυνατότητε πέραν των βιοκαυσίμων. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα καυσίμα που χρησιμοποιούμε στον τομέα των μεταφορών, τα βιοκαύσιμα αυτά θα πρέπει να μας επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε τις εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, να μην επιβαρύνουν την αποψήλωση και τις τιμές των τροφίμων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιέσει για την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων και όπως είπα και για τι ανανεώσιμε πηγέ της μεταφορέ και για τα ηλεκτροκινητά οχήματα. Επίσης, το όριο του 5% πιστεύω ότι είναι υπερβολικά υψηλό. Πρέπει να μην ξεπεράσουμε το 4%. Η μείωση του ορίου στο 5% δεν θα μα επιτρέψει να επιδιώξουμε τους στόχους αεφορία που προανέφερα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, εύληπτου στόχους και για τα κάψιμα δεύτερη γενιάς. Θα πρέπει να είναι δεσμευτικός αυτός ο στόχος, τουλάχιστον στο 2%. Ε, ίσως και παραπάνω, αλλά τουλάχιστον 2%. Έπειτα θα πρέπει στην αγορά σήμερα να διατίθενται τέτοια προϊόντα. Βλέπουμε την εθανόλη δεύτερη γενιά, που είναι πολύ σημαντική ε, και από την σκοπιά της παραγωγής. Πολλοί είναι εκείνοι που ρωτούν αν έχουμε πρώτες ύλε για δεύτερη γενιά καύσιμα και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι έχει υποπροϊόντα διαθέσιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λόγω χάρη τα άχυρα. Και αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή δεύτερης γενιάς εθανόλης. Τον Ιανουάριο του 2012 το Bloomberg Finance δημοσίευσε μια έκθεση για το δυναμικό ε, δημιουργία της εργασία στον κλάδο των καυσίμων δεύτερης γενιάς. Εδώ πραγματικά νομίζω ότι πολλές θέσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε και η έκθεση αυτή το διαβεβαιώνει. εκατό 100.000 θέσεις εργασίας εάν προσθέσουμε στην παραγωγή της βενζίνης με δεύτερης γενιάς εθανόλης. Βεβαίως θα υπάρξουν και παραπροϊόντα αλλά μπορούμε να διαβεβαιωθούμε και γι' αυτό, να λάβουμε μέτρα και γι' αυτό χωρίς να βλάψουμε το περιβάλλον. Μπορούμε να δημιουργήσουμε 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2030 και βεβαίως να έχουμε κατά νου και τους ε, παράπλευρους παράγοντες. Ευχαριστώ ο κύριος Τούρμες για τρία λεπτά. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Τούρμες. Ευχαριστώ για την συνεισφορά σας. Αυτό που μας πρότεινε ο Επίτροπος δυστυχώς έχει έρθει με μια καθυστέρηση δύο ετών. με τις διαπραγματεύσεις για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Το Δεκέμβριο του 2008 ήδη τα ζητούσαμε αυτά και ξέραμε ότι η πρώτη γενιά βιοκαυσίμων ή τέλο πάντων γεωργικών καυσίμων θα δημιουργούσαν προβλήματα το μόνο που καταφέραμε τότε είναι να διαβεβαιώσουμε ότι η αποτίμηση κύκλου ζωή για τα δύο κάψιμα θα είναι ολοκληρωμένη και όχι μόνο, δεν θα λαμβάνει μόνο υπόψη την, χρήση, την πρωτογενή χρήση της γης. Τελικά το καταφέραμε, αλλά νομίζω καλό είναι που τώρα έρθε με αριθμητικά στοιχεία μας εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν οι Ηνωμένε σχετική νομοθεσία παρόλα αυτά και δεν είναι δική μα αποκλειστικότητα. Θα μπορούσαμε να βασιστούμε στην εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που πρέπει πάντως να κάνουμε είναι να δούμε ότι οι πολιτικές αυτές δεν είναι απλώς ε, πολιτικές εντολής και εκτέλεσης. Θα πρέπει να δώσουμε ισχυρές ενδείξεις και προς την αγορά. Και αυτό θα γίνει εάν τα συμπεριλάβουμε αυτά στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Μόνον έτσι οι εταιρείε δίληση θα έχουν κίνητρο για να επιδιώξουν υψηλότερου στόχου καταπολέμηση των ε, ε, εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα και θα παράγουν τέτοια βιοκαύσιμα. Εάν δεν το συσχετίσουμε αυτό με την πραγματικότητα των τιμών στι αγορέ, Πάλι σχεδιάζουμε μια πολιτική εντολής και εκτέλεσης. Λε και είναι κάτι το αυτόματο. Όχι, πρέπει να βρούμε έναν ευθύ τρόπο. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίε να θίξουμε τέτοια σημεία και θα το κάνω αυτό. Σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά για την όλη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Βίνταλ Κουάντρας για την ε, ξεκάθαρη αυτή η παρουσίαση του πόσο πολλές δυσκολίε έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ και να τον στηρίξω και εγώ από την πλευρά μου για την ε, κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει. Να παρατηρήσω ότι προφανώς χρειαζόμαστε σαφήνεια για το θέμα αυτό, προκειμένου να τονώσουμε τις επενδύσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ε, σχεδόν ε, μισό δις στερλίνες επενδύσεις σε συγκεκριμένες υποδομές και εργοστάσια και θέλουν να δουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε εμείς. Εγώ αυτό που ρωτώ πάντω είναι αυτό το 10% ηλεκτροκίνητων οχημάτων από πού θα προκύψει για να επιδιώξουμε αυτό το στόχο. Διότι εδώ συμφωνώ με τον κύριο Βίνταλ Κουάντρα. Δεν θα γίνει όπω το έχουμε φανταστεί. Έπειτα. Α γινόταν μια μελέτη αντικτύπου Ας είχαμε και λίγο φως στην όλη υπόθεση. Διότι γύρω-γύρω γυρνάμε από το ίδιο θέμα με τα βιοκαύσιμα. Ωραίο είναι, μας αρέσει, αλλά μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν και μειονεκτήματα και δεν είναι και τόσο απλό να εφαρμοστεί ως λύση. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που πρέπει να τα ξανασκεφτούμε. Βέβαια αυτή είναι μια διερευνητική συζήτηση και πρέπει να ξανευχαριστήσω τον κύριο Βίνταλ Κουάντρας που πραγματικά ανέλαβε αυτό το έργο που είναι γεμάτο προκλήσει, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον βοηθήσω από την πλευρά μου. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Αφού ακούσαμε τον εισηγητή μα και του κοιόδη εισηγητέ, θα παρακαλέσω την κυρία Λεπάζ, ε, την εισηγητρία τη ΕΜΒΗ, να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Βινταλ Κουάντρας, με τον οποίο θα έχω τη χαρά να συνεργαστώ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και αυτό για ένα θέμα που δεν είναι καθόλου απλό. Εδώ συμμερίζομαι πλήρως τις παρατηρήσεις του για την δυσκολία του όλου εγχειρήματο. Νομίζω είναι πολλά τα σημεία όπου σχετικά άνετα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Το πρώτο, ως στόχος μείωσης και συμβολή στη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου είναι σίγουρος. Αυτό θα πρέπει να είναι η πηξίδα μας ως προς τον προσανατολισμό που θα ακολουθήσουμε. Δεύτερο σημείο, δεύτερο στόχος. Ο στόχος να λάβουμε υπόψη τις επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει από όλους τους ε, ενδιαφερόμενους και ε, δραστηριοποιούμενους σε αυτόν τον τομέα. Έχουν επενδύσει κάποιοι στα δύο κάψιμα της πρώτης γενιάς και μάλιστα έτσι που κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης δεν μπορούμε να τους πλήξουμε ούτε ως προς την ε, ε, απασχόληση ούτε προς τις θέσεις εργασίας. Τρίτη παρατήρηση, πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα για τον προσανατολισμό που θέλουμε να λάβει αυτή η πολιτική. Πρώτο στοιχείο δεν είναι αηφόρος ο συλλογισμός, δεν εξυπηρετεί την αηφορία, αν πρέπει να σκεφτούμε το να επιλέξουμε μεταξύ του να τρώμε ή να οδηγούμε. Ξέρουμε ποιο είναι το παγκόσμιο σκηνικό ε, και μάλιστα από καιρό. Συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει είναι να δώσουμε κάποιο νέο μήνυμα. Δεν μπορεί να είναι και ρηξικέλευθο, διότι από την οδηγία του 2009 και από τις συζητήσεις που είχαν γίνει στο Κοινοβούλιο τότε, τα σημεία αυτά είχαν προκύψει. Τα είχαμε θίξει. Είχαμε πει ότι πρέπει να περάσουμε στα γεωργικά καύσιμα τη δεύτερη γενιά. Η ανάγκη αυτή είχε τονιστεί ακριβώ διότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα αηφόρο, βιώσιμο, όταν στις χώρες του Νότου, αλλά όχι μόνον, χρησιμοποιούνται τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα για να μετατραπούν σε βιολογικά καύσιμα. Αυτό τα αποστερεί από ένα μέρος των πολιτών, από ένα μερίδιο του πληθυσμού. Τους είναι αναγκαίο όμως για την επιβίωσή τους στην καθημερινότητα. Νομίζω σε αυτά τα στοιχεία όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε. Έπειτα το θέμα είναι πώς θα βρούμε το σωστό επίπεδο, το σωστό βαθμό. Και θα είναι τα ποσοστά 5% θα είναι πρότυπο κανόνα, προδιαγραφή. Πρέπει να έχει ένα σαφή προσανατολισμό η οδηγία, να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Πρέπει ή δεν πρέπει να διακρίνουμε την εθανόλη από το βιοντίζελ. Οι επιπτώσεις από την πλευρά του ILOG δεν είναι καθόλου ίδιε ίδιες για αυτά τα δύο κάψιμα. Έπειτα, πρέπει ή δεν πρέπει να διατηρήσουμε τους παράγοντες που ε, προτείνει η Επιτροπή και βάσει ποιων κριτηρίων. Δεδομένου ότι το όλο θέμα με αυτή την οδηγία, και θα συμφωνήσω εδώ με όσα είπε προλίγου ο συνάδελφος, θα πρέπει να αναπτύξουμε νέα τεχνολογικά μέσα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας με τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Σαφή μηνύματα χρειάζονται λοιπόν και για τις επενδύσεις και για την βιωσιμότητα, ώστε να υπάρχει συνέχεια στις επενδύσεις που θα γίνονται. Έπειτα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους παράγοντες Άιλο και όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Βιντάλ Κουάντρας, θα πρέπει να τους αναθεωρούμε διαρκώς, συστηματικά, διότι θα προχωρούν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτή βεβαίω είναι μια καλή κατεύθυνση, ασχέτως με το αν πρέπει να είναι η προσέγγιση σφαιρική ούτε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε να ευνοήσουμε τα βιολογικά καύσιμα, των οποίων οι συνέπειε μακροπρόθεσμα θα είναι αρνητικέ και όχι θετικέ σε σχέση με του συνολικού μα στόχου. Δηλαδή, καταπολέμηση των, των απομπών αερίων, ε, αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή είναι, κυρία Πρόεδρε, γενικώ η στάση μα ω προ την σύνταξη τη έκθεση αυτή. Πραγματικά ο παράγον ILOG θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, είναι κάτι ε, ιδιαίτερα σημαντικό και θα ήθελα να εντοπίσουμε τον σωστό βαθμό, ώστε οι επενδυτές μας να ε, αισθάνονται ασφάλεια και επίσης να υπάρχει ένας δυναμικό ρυθμό στις επενδύσεις που θα γίνονται. Και να έχουμε ορθολογικά κριτήρια. Δύσκολο μεν, αλλά γίνεται. Να κάνουμε όσο το δυνατόν τις καλύτερες επιλογές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Λέπαζ. Και τώρα ο κύριο Γκριμπς. Ε, <coughs> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Βιδάλ Κουάντρας. Συμφωνώ, το ερώτημα είναι θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το 10% ανανεώσιμων στις μεταφορές Θέλουμε επίση να δώσουμε κίνητρα εις τους ε, επενδυτέ για το μέλλον και επομένω να δούμε το πώς θα υπάρξει κάποιο είδου εμπιστοσύνη που την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε. Να σας πω το παράδειγμα από την Πολωνία. Ε, στην Ευρώπη παράγουμε βιοδίζελ και στη ΣΕΙΠΑ αλλά και στη Λατινική Αμερική μόνο βιοεθανόλια. Ή στην Πολωνία χρειαζόμαστε 1,2 εκατομμύρια τόνους ελαιοκράμβες, τέλος πάντων ε, ελαιοκράμβες, για να παραγάγουμε το, το αντίστοιχο. Μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια τόνους και παράγουμε 3 εκατομμύρια ε, από τα 3,5. Οτιδήποτε πάνω από 1,2 εκατομμύρια τόνους μέχρι τα 3,5 εκατομμύρια ε, είναι η διαφορά από την παραγωγή και είχαμε το κινήτρο το οποίο μας βοήθησε σε σχέση με τις με τα κίνητρα τα οποία δόθηκαν για, τα, ε, για αυτά τα τα, τα, τα, τα, για, αυτές, τις, ε, τις καλλιέργειες και τελικά όμως ο ιδιωτικός τομέας έδωσε τα κίνητρα. Βεβαίως και χρειάζεται μακρόπνοη επένδυση. Επομένω, τώρα πού το πάτε. Τι, τι προβλήμα θα ξεπεταχτεί αύριο. θα είναι ο της ΓΕΕΣ. Τώρα μας λέτε για περιορισμό του στόχου στο 5%. Μάλλον θα πρέπει να κάτσουμε και να θεωρήσουμε αυτό το οποίο τώρα ε, πάμε να κάνουμε. Καταλαβαίνουμε ποια είναι τα αποτελέσματα από τη χρήση του παράγοντα ILOP και νομίζω φυσικά θα πρέπει να επιλέξουμε με τρόπο υπεύθυνο, αλλά δεν θα πρέπει να καταρακώσουμε την εμπιστοσύνη γιατί αυτό θα γίνει όταν κανείς αλλάζει το πλαίσιο, το ρυθμιστικό κάθε χρόνο. Σκεφτείτε επομένως τι είναι το πιο σημαντικό από πλευράς γεωργίας. 80-70% του συνόλου των καλλιεργιών είναι σίτερα Και σε πολλές χώρες. Έχουμε πατάτες, έχουμε επίσης και ε, κοκκινοβούλια Οπότε έχουμε αυτή τη συγκυκλική εναλλαγή και δεν είναι δυνατόν να γίνει κανένα είδου ε, αλλαγή σε αυτή τη σειρά. Το βιοντίζελ και η βιοεθανόλη ως παραγωγή, ξέρετε, οδηγούν σε κάποιους 780 τόνους ε, που παράγονται ε, ως κτηνοτροφή. Δεν είναι αυτό το επιλέγουμε σε κύριε Λαπάζ. Δεν ισχύει το ότι όταν γίνεται αυτή η παραγωγή είναι σαν να κόβουμε το φαγητό. Γιατί εμείς ε, εισάγουμε πάρα πολλά τροποποιημένα γενετικά σιτηρά αντί να παραγάγουμε κάποιο είδου υψηλή πρωτενη σε Άρα για πολλού λόγου θα πρέπει να δούμε το ζήτημα με κάποια οπτική γωνία που έχει τα πνεύματος. Να μην τα βλέπουμε πάρα πολύ στενά μυαλά όσον αφορά τα καύσιμα αυτά τα δύο καύσιμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχει προχωρήσει η ώρα θα είμαι σύντομη μετά και τον πρώτο γύρο συζήτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Βιδάλ Κουάντρας. Συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες και θέλω μόνο να πω πως ε, δεν πρέπει να καταστρέψουμε την εμπιστοσύνη που υπάρχει εδώ πέρα και να υπάρξει και μία εγγύηση των ε, επενδύσεων. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε τα βιοκαύσιμα της ε, πρώτης γενιάς και μετά να λέμε χι ε, και να καταστρέφουμε ακριβώς την εμπιστοσύνη των ε, μεσαίων επιχειρήσεων που έκαναν επενδύσεις και εξαρτώνται για την ύπαρξή τους τώρα. Ε, για να παραμείνουν στην αγορά βιοκαυσίμων. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τα βιοκαύσιμα της ε, δεύτερης ε, γενιάς. Και υπάρχει, αν θέλετε, μια κάποια επιτυχία εδώ πέρα για... και πρέπει να βοηθήσουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν το βιοκαύσιμα αυτά της ε, πρώτης γενιάς. Και ευχαριστώ τον κ. Βιδαλκόντρας γιατί ανέπτυξε τα διλήμματα που υπάρχουν και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα γενευτεί η μεταβολή. Σας ευχαριστώ η Κομισιόν αν θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όντως, έχει περάσει ώρα, οπότε και εγώ θα είμαι σύντομος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη συζήτηση. Θεωρούμε ότι αυτά τα τρία ζητήματα κλειδιά τα οποία ανέφερε ο εισηγητής είναι πάρα πολύ εύστοχα. Αυτό το 5% το, το η πολλαπλή, ο και ακριβώς τώρα αυτά και συζητούμε με το Συμβούλιο. Ακριβώς, ακριβώς αυτά θα συζητήσουμε. Τώρα, από πλευράς δικής μας. Θεωρούμε ότι η πρόταση που έχουμε διατυπώσει είναι η σωστή απόκριση σε αυτέ τις προκλήσεις που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα ξέρουμε πολύ περισσότερο το 2008 τότε που άρχισε να διαμορφώνεται αυτή η οδηγία με τη διαπραγματεύση. Και επίση ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλά θέματα στον αφορά αυτέ τι έμεσε εκπομπέ και οπότε και θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε κατά τον βητά τρόπο και θεωρούμε ότι η πρόταση εδώ αυτή ε, αποτελεί τη, τη, τη σωστή εξορροπήση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων. Δηλαδή, έτσι, μειώνονται αυτέ οι έμεσε ε, εκπομπές και ταυτόχρονα όμως λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσει που ήδη έχουν τελεστεί. Όμως το πιο σημαντικό από όλα είναι το ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα το οποίο έτσι στέλνουμε σε σχέση με το ποιο είδους βιοκαύσιμα θέλουμε για το μέλλον. Και αυτό επίσης το ανέφεραν κάποιοι από τους αγορητέ σήμερα. Δηλαδή Τώρα διψάγει ένα τέτοιο μήνυμα η βιομηχανία και επίση θα πρέπει να το στείλουμε. Και επίση θα πρέπει να δούμε τι θα πούμε γιατί θέλουμε να μειώσουμε για ε, τα βιοκαύσιμα πρώτη γενιά, αυτά τα οποία έχουν τι πιο πολλέ εκπομπέ, να δώσουμε κάποια αντικίνητρα. Όμω να δώσουμε παραπάνω κίνητρα μέσω αυτού του τετραπλού συνυπολογισμού και να το συζητήσουμε αυτό από δύο όχι. Αλλά έτσι τουλάχιστον εντοπίζουμε εκείνα τα βιοκαύσιμα τα οποία είναι σήμερα τα πιο σημαντικά. Τέλο πάντων, νομίζω ότι έχουμε βρει τη σωστή ισορροπία και θα ήθελα να σας πω ακριβώς το τι γίνεται όσον αφορά την ε, μελέτη των επιπτώσεων και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι ό,τι λίγο μου θα έχει την ευκαιρία να τα μελετήσετε. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεισφορά τη Ο λόγος για τα συμπεράσματά του στον κύριο Βιντάρ Κουάντρας. Sí, muchas gracias. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμεθα ή ικανοποιημένοι μετά από αυτήν την ε, ανταλλαγή απόψεων, μετά από αυτή την πρώτη συζήτηση. Διότι νομίζω καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι μπορέσαμε να οριοθετήσουμε και να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να εξεύρουμε λύση. Λύση που θα συγκεντρώνει τις απόψεις πλειοψηφίας. Σήμερα όμως διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κοινά σημεία συμφωνίας, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να ε, ε, δεν θέσουμε κινδύνο τις ήδη τελεστήσεις επενδύσεις. Θα πρέπει να τις ε, προστατεύσουμε. Επίσης, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί εντύπωση ότι η νομοθεσία είναι ασταθής και απρόβλητη. Γιατί και αυτό κάνει κακό στις επενδύσεις και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητος που και αυτό για τον κλάδο θα είναι πάρα πολύ για το μέλλον του. Επίσης, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δούμε το πώς θα περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της έμεσης αλλαγής της χρήσης της γης. Πώς θα γίνει αυτό. Εδώ θα πρέπει να κάτσουμε και να συμφωνήσουμε. Πρότεινε κάποιο πράγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 5% Έχουμε αυτή την λίστα με τα δύο καύσιμα Δευτέρας και Τρίτης Γενέας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να τύχουν πριμοδότησης όσον αφορά το ότι συμβάλλουν ή στον στόχο. Έχουμε, έχουμε λύσεις. Ας τις μελετήσουμε και ως συνήθως ας ε, έχουμε ως βάση το αξιόλογο έργο της Επιτροπής και να το βελτιώσουμε περισσότερο. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Περιμένω λοιπόν και υπολογίζω εις την, την κρίση και στην βοήθεια όλων των συναδελφών. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βιντάλ Κουάντρα. Επόμενη συζήτηση για το θέμα αυτό στις 24-25 Απριλίου. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους. Να θυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 24-25 Απριλίου. Αυτή της 11 Απριλίου ακυρώθηκε. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την ε, μέρα δουλειάς που περάσατε μαζί μου. Καλώς σας βράδυ.